Καλησπέρα σε όλους. Ε, ξεκινάμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Σημείο 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Για τεχνικούς λόγους, η διερμηνία δεν είναι εγγυημένη σε όλες τις γλώσσες. Η γλώσσα που λείπει σήμερα είναι τα λιθουανικά. Σημείο 2 της ημέρης διάταξης. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 12ης Δεκεμβρίου και της 19ης και 20ης Δεκεμβρίου. Και εδώ, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων εγκρίνονται. Να σας ενημερώσω επίσης ότι η σημερινή συνεδρίαση αναμεταδίδεται στο webstream, μέσω του webstream. Ωραία λοιπόν, ξεκινάμε με το σημείο 4. Εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των ε, προβάτων. Η συγγετής είναι ο κ. Βοζιγόφσκι. Έγκριση του σχεδίου σύστασης για δεύτερη ανάγνωση. Ξεκινάμε τις ψηφοφορίες, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρώτη ψηφοφορία είναι η θέση της δεύτερης ανάγνωσης όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων. Στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής εξετάσαμε το σχέδιο σύστασης του κυρίου Βοζιγουόφσκι για να υιοθετήσουμε τη θέση σε πρώτη ανάγνωση ε, χωρίς τροποποίησης. Καμία τροπολογία δεν υποβλήθηκε σε αυτό το σχέδιο σύστασης. Γι' αυτό προτείνω να περάσουμε αμέσω στην ψηφοφορία. Καταρχήν σα ρωτώ αν έχετε όλοι τι κάρτε τη ψηφοφορία. Έχετε τι κάρτε σα όλοι. Ωραία. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε. Βοσιγόφσκι, θες το λόγο? Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε αμέσω τότε. Και favorevole. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Όχι. Ωραία. Εγκρίνεται. Okay. Bene. Avanti. Andiamo al punto 5. Περνάμε στο σημείο 5. Distribuzione di generi alimentari. Διανομή τροφίμων υπέρ των ενδεέστερων. Εισηγητής ο Πρόεδρο Σικέρσκι. Περνάμε στην έγκριση του σχεδίου σύσταση για δεύτερη ανάγνωση για το πρόγραμμα διανομή τροφίμων στου ενδέστερου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση του Συμβουλίου θετήθηκε στι 23 Ιανουαρίου και ανακοινώθηκε επισήμω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στι 2 Φεβρουαρίου. Η θέση του Συμβουλίου προβλέπει το σημερινό πρόγραμμα να ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2012 και να συνεχιστεί μέχρι το 2013. Επίσης, η Κομισιόν έχει διαβιβάσει σε κατ' εφαρμογή του άρθρου 254 της Συνθήκης μια ανακοίνωση σε σχέση με τη θέση του Συμβουλίου που διανεμήθηκε σε όλους σας υποστηρίζει το αποτέλεσμα των διοργανικών διαπραγματεύσεων και δέχεται την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση με στόχο να εγγυηθεί τη συνέχιση του καθεστώτος μέχρι το 2013. Σε ένα παράρτημα της σημερινής ανακοίνωσης, αυτής της ανακοίνωσης η Κομισιόν κάνει και μια δήλωση. Πιστεύω ότι μετά την υιοθέτηση αυτού του φαγγέλου στην Ολομέλεια που προβλέπεται για την επόμενη εβδομάδα θα ήταν σκόπιμο να επανέλθουμε και να εκφραστούμε για αυτές τις δηλώσεις σε μία από τις επόμενες ολομέλειες. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε λοιπόν τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματο, νομοθετικού ψηφίσματος. Και ζητώ από τον ε, Αντιπρόεδρο Σικέρης και αν θέλει να πάρει το λόγο. Αν όχι δεν θέλει. Α, όχι θέλει. Τα όσα έπρεπε να υποθούν υπόθηκαν κύριε Πρόεδρε, οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας παρακαλέσω να το εγκρίνουμε χωρίς καμία αλλαγή ή τροποποίηση. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κύριε Σικέρσκι, θυμίζω... Όχι, δεν χρειάζεται. Μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Σικέρσκι και σας ευχαριστώ όλους. Περνάει από την Ολομέλεια στο επόμενο Στρασβούργο. Σημείο 6. Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο, στρατηγική της ΕΕ για τη βιοπικιλότητα, η συγγήτρια είναι η κυρία Βασίλικα Βιόρικα Ντάντζιλα. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στην παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης ε, για την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Στρατηγική 2020 για τη Βιοπικιλότητα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το ρόλο της γεωργίας και το αντίκτυπο της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, στην βιοεπικιλότητα. Σημειώνουμε ότι το σχέδιο έκθεσης, το οποίο εκπονήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβάνει την πρόταση αύξησης του ποσοστού άμεσων πληρωμών που θα έπρεπε να είναι αφιερωμένη στο, στις περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, το περίφημο 7%. Πιστεύω πως αξίζει να κάνουμε μια προσεκτική αξιολόγηση εμείς, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτές οι άμεσες πληρωμές, για τις οποίες η δική μας Επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια. Και τώρα, αγαπητή Βασιλική, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η διατήρηση της βιοπικιλότητας ε, έχει πλέον καταστεί τόσο ευρωπαϊκή όσο και διεθνή προτεραιότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Ορισμένοι αρνούνται ότι υπάρχει κίνδυνο εξαφάνιση ειδών, αλλά οι επιστήμονε αφιστούν την προσοχή μα σε ένα ε, πάρα πολύ σοβαρό φαινόμενο όπω αυτό. Βέβαια δεν θα πρέπει οι προσπάθειε για τη διατήρηση τη βιοπικιλότητα να περιορίζονται σε ορισμένα και μόνο οικοσυστήματα, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε την υποβάθμιση οποιονδήποτε οικοσυστημάτων, όπου και αν είναι αυτά. Ε, δεν πρέπει επίσης και τα δασικά οικοσυστήματα να τα παραγνωρίζουμε γιατί παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και για τη βιοπικιλότητα αλλά και για τη διατήρηση της ισορροπίας ε, του γεωλικού συστήματος. Ε, η φυσική κληρονομιά είναι και πολύ σημαντική οικολογική κληρονομιά που συμβάλλει στην ευημερία της ανθρωπότητας. Επομένως, θεωρώ ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να αξιοποιήσουν καλύτερα τους φυσικούς πόρους και να περιορίσουν την υποβάθμιση της βιοπικιλότητας. Όταν μιλάμε για βιοπικιλότητα, πρέπει να σκεφτόμαστε επίσης ε, τα φυσικά πάρκα που είναι υποπροστασία ή θα περιληφθούν στον κατάλογο των προστατευόμενων ε, φυσικών ε, πάρκων, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και την λειτουργική βιοπικιλότητα. Η λειτουργική βιοπικιλότητα διαδραματίζει ένα ρόλο ώστε να διατηρηθεί η πανίδα, ιδίω τα έντομα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την επικονία των φυτών. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαιρετίζουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν μέτρα σε σχέση και με τον πρώτο και με τον δεύτερο πυλώνα και τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της βιοπικιλότητας. Σε αυτά τα μέτρα θα πρέπει να συσχετίσουμε και οικονομικούς δείκτες έτσι ώστε να είναι βιώσιμοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την εκπεριτροπής καλλιέργεια, τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών. Θα πρέπει δε να ενθαρρυνθούν και οι καλλιέργειες οι οποίες ε, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευρά τη βιοπικιλότητας. Για παράδειγμα, καλλιέργειες που βοηθούν τη φυσική επικονίαση. Γύρω στα 20 δις είναι το ποσό που θα πρέπει να δετεθεί για να υπεξασφαλίσει η διαδικασία της επικονίασης. Είναι πολύ σημαντικό να αναλυφθεί δράση υπέρ της βιοπικιλότητας. και σε ε, δημόσια πάρκα, κοντά σε σιδηροδρόμους, ε, ε, στα περίχωρα των αστικών κέντρων, μεταξύ άλλων. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ενταχθούν σε προγράμματα χωροτεξικού σχεδιασμού. Η διατήρηση των φυσικών πόρων, των γενετικών, φυσικών, ζωικών πόρων, οι αγροτεχνολογικές διαδικασίες, όλα αυτά είναι απαραίτητα ώστε να εξασφαλιστούν οι ανάγκες των ε, μελλοντικών γενναιών. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και αποτελεσματική συνεργασία σε ό,τι αφορά τους γενετικούς, ζωικούς και φυτικούς πόρους. Θα πρέπει να διατηρηθούν οι πόροι αυτοί και θα πρέπει να ευνοηθεί η προσαρμογή τους ε, στην αλλαγή του κλίματος. Θα πρέπει επίσης να εναρμονιστούν και οι δράσεις σε εθνικό, τοπικό, περιφερειακό επίπεδο και να υπάρξει συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Δεν θα πρέπει να λεξιτοποιήσουμε το ρόλο της γεωργικής έρευνας, ούτε και το ρόλο της τεχνολογικής καινοτομίας. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη βιοπικιλότητα και των σχεδίων ανάπτυξης υπαίθρα των κρατών μελών. Έτσι ε, θα επιτευχθεί ο στόχος της ε, διατήρησης βιοπικιλότητας. Οι αγροτικές περιοχές θα πρέπει και αυτές να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν ώστε να αναπτυχθεί και η βιοπικιλότητα. Προς εκπλήρωση των στόχων αυτών η Ευρώπη πρέπει να βάλει τη βιοπικιλότητα στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της. Επίσης θα πρέπει να γίνει και, μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του πληθυσμού. Οι νέες γενιές ε, θα πρέπει να παροτρινθούν ε, ώστε να ανακαλύψουν τη φύση. Πρέπει να στηρίξουμε τις ε, πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών υπέρ της βιοποικιλότητας. Θα πρέπει να προωθήσουμε, να ενισχύσουμε και την προσπάθεια που κάνουν οι θελοντικές οικολογικές οργανώσεις να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καλές πρακτικές που θα πρέπει και να γίνουν γνωστέ χάρη στι εκστρατείε ευαισθητοποίησης τη οποίες μίλησα. Οι εκστρατείε αυτέ θα πρέπει να στοχεύουν σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, σε όλους τους πολίτες. Νομίζω ότι τα προγράμματα επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση θα πρέπει επίση να προσαρμοστούν, ιδίω ό,τι αφορά την ε, κατάρτιση στο Γεωργία και στου συναφεί τομεί. Για να δοθεί έμφαση στη βιοπικιλότητα, πρέπει ε, να αναπτυχθούν οι σχετικέ δεξιότητε στην Ευρώπη και να υπάρξει να παρασχεθεί σχετική εκπαίδευση. Θα πρέπει επίση να ενθαρρύνουμε τα τοπικά περιφερειακά σχέδια, καθώς και τα διασυνοριακά σχέδια για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη μη κυβερνητικών οργανώσεων και θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και με τον πανεπιστημιακό κόσμο όλα αυτά τα θέματα ή άλλως απασχολούν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, άρα θα πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια εφαρμογής ε, της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοπικιλότητα. Προσπάθησα να σας εκθέσω εν συντομία τα θέματα που αναφέρω και στην γνωμοδότησή μου και περιμένω τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας σε σχέση με αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα της βιοπικιλότητας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε κυρία Ντάνσιλα. Σε ευχαριστούμε Βασιλική και τώρα ξεκινάμε τη συζήτηση. Έχουν εγγραφεί διάφοροι συνάδελφοι και ξεκινάμε με τον κύριο Ρέιμερς. Την κυρία Ρέιμερς, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ποικιλότητα είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για το μέλλον μας. Όταν όμως το συζητούμε θα πρέπει να αποφύγουμε να προσεγγίζουμε το πρόβλημα μόνο από την οπτική της γεωργίας ή των ε, περιοχών της υπαίθρου. Θα πρέπει επίσης στις πόλεις ε, ή ε, στις πυκνοκατοικημένες περιοχές να εφαρμόζουμε αυτήν την στρατηγική. Πρέπει επίσης να φροντίσουμε, να προσέξουμε, ώστε στο πλαίσιο της κοινή γεωρικής πολιτικής ε, υπάρχουν προγράμματα που λειτουργούν πολύ σωστά στο δεύτερο πυλώνα, που λειτουργούν θετικά για τη βιοπικιλότητα. Θα πρέπει να αποφύγουμε να τα αμφισβητήσουμε. Και, να... και θα πρέπει να φροντίσουμε στον ε, δεύτερο πυλώνα ε, να έχουμε ένα καλό μοντέλο, όχι αυτό που τώρα πια δεν λειτουργεί Ευχαριστώ. πολύ. Θα πρέπει να πω ότι βρίσκω πολύ καλή την έκθεση του συναδέρφου και νομίζω ότι η προσέγγιση που επέλεξε ε, το ότι παίζει και στην γεωργική πολιτική βιοποικιλότητα πολύ σημαντικό ρόλο είναι μια προσέγγιση που αξίζει να στηρίξουμε. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω κατά της ιδέας ε, να υπονομεύσουμε το 7% με τρόπους, με στρατηγικές που τελικά ε, θα οδηγήσει στο να μην συζητιέται πια αυτό το 7% στον πρώτο πυλώνα. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ε, έχουν να προσφέρουν οι εκμεταλλευσει. Αρκετέ βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο. Πολλέ ε, συμμετέχουν στα μέτρα τα γεωργικά και περιβαλλοντικά ενώ άλλες δεν το κάνουν. Θα πρέπει, νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον η βιοπικιλότητα να εντάσσεται και στον πρώτο πυλώνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τώρα το λόγο έχει ο Μάρτιν Όσλιν και μετά η Ελίζα Μπατιγέγκλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η γεωργία, σε αντίθεση με, πολλές, με πολλούς άλλους τομείς, έχει ε, βασική ευθύνη για τη ε, διασφάλιση της βιοποικιλότητας. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Ε, αποτελεί και αιτία για την απώλεια βιοπικιλότητας. Ε, γι' αυτό ε, είναι σωστό στην γεωργική πολιτική να κάνουμε κάτι για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Οι προτάσεις της Κομισιόν θα πρέπει να εξετεστούν περαιτέρω σε πολλά σημεία αποτελούν τον κατάλληλο δρόμο ώστε να καταπολεμήσουμε την απώλεια της βιοπικιλότητας. Η κυρία Ρόντουστε ήδη αναφέρθηκε στο 7% θα πρέπει αυτό το μέτρο να εντάσσεται στον πρώτο πυλώνα, όχι στον δεύτερο. Σε περιφέρειες όπου, υπάρχει, ε, όπου διατηρείται η βιοπικιλότητα δεν ε, χρειάζεται να ενισχύσουμε τα μέτρα. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε τα μέτρα ε, σε τομείς που έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Γι' αυτό σωστό είναι στον πρώτο πυλώνα να συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα αυτά. Αυτό ε, δεν σημαίνει ότι ε, χρειάζεται να παραιτηθούμε από ενισχυτικά μέτρα στον ε, δεύτερο πυλώνα. Επίσης, θέλουμε να διατηρήσουμε και ε, κάποια γεωργικά φυτά. Αυτό μπορεί να μην ε, αναφέρεται στην πρόταση της Κομισιόν, αλλά έχουμε χάσει πολλά είδη ε, και θα πρέπει να κάνουμε κάτι εδώ. για παράδειγμα, έχουμε σημαντική απώλεια γενετικών πόρων στα όσπρια. Τελικά, το θέμα δεν είναι μόνο να προστατεύσουμε την ε, φύση, αλλά είναι και οικονομικό, διότι με την απώλεια γενετικών πόρων ε, Έχουμε και οικονομική απώλεια, μπορούμε να την εκφράσουμε σε ευρώ. Είναι λοιπόν προ όφελο όλων να διατηρήσουμε τους πόρου αυτούς και να τους αναπτύξουμε περαιτέρω. Γι' αυτό θα ήθελα στην έκθεση αυτή ε, να δω περισσότερα για την ε, κοινή ε, γεωργική πολιτική. Να επικεντρώσουμε την κοινή γεωργική πολιτική στην τήρηση της στρατηγικής. Αυτό έχει να κάνει και με την αξιοπιστία μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τρίτες χώρες να διατηρούν και να προστατεύουν τη βιοπικιλότητά τους, ενώ εμείς εδώ στην Ευρώπη εδώ και χρόνια να μην μπορούμε να πετύχουμε τους αντίστοιχους στόχους μας. Πρόκειται λοιπόν για δύο καθυστερημένες ε, προτάσεις. Ε, θα πρέπει να διατηρήσουμε την βιοπικιλότητα στα ε, τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάρτιν, η Ελίζαπετ Γέγκλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τις εξηγήσεις που μας έδωσε για αυτό το αδιαμφισβήτητα σημαντικό θέμα. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν, ωστόσο να τονίσω ότι είναι σημαντικό θέμα. Είναι ένα θέμα το με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε τατικά κατά τις ε, διαπραγματεύσεις για την κοινή γεωργική πολιτική. Δεν θα ήθελα να προδικάσω τη θέση μας ώστε ε, να δυσκολευτούμε μετά να οπισθοδρομήσουμε. Θα υποβάλω τροπολογίες οι οποίες ε, κυρίως θα στοχεύουν στις προσπάθειές μας στις περιφέρειες, ώστε να μπορούμε να αυξήσουμε την βιοπικιλότητα. Η θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι δεν είναι όλα κακά αυτά που κάνουμε στην, ε, στον τομέα τη Γεωργία. Υπάρχουν και καλά στοιχεία και θα πρέπει να σκεφτούμε ε, σε όλη την Ευρώπη, στον πρώτο πυλώνα δηλαδή και επιπλέον στον δεύτερο πυλώνα στι διάφορε περιφέρειες να κάνουμε περισσότερα από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αν ε, επιχειρηματολογήσουμε σωστά θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε σημαντικά στις συζητήσεις για την κοινή γεωργική πολιτική και αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχο μας. Ευχαριστώ, Ελίζαμπετ. Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος Πόλσον και μετά ο Αλμπερτές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν συζητάμε την βιοπικιλότητα να θυμόμαστε αυτό το απλό γεγονός ότι η γεωργία τα δάση και εν μέρη η αλληλεία ε, διαχειρίζονται τους φυσικούς μας πόρους. Στο παρελθόν πάντα λέγαμε ότι θα πρέπει να ε, προστατεύσουμε ευαίσθητες περιοχές ε, και αυτό συνεχίζει να ισχύει. Αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε ότι Πρέπει να έχουμε οικολογικούς διαδρόμους στην Ήπεθρο και, στην, ε, και στις γεωργικές περιοχές και στις ε, ε, περιοχές εντατικής δασοκομείας, ώστε όλοι οι οργανισμοί Όλοι, όλοι οι γενετικοί πόροι θα πρέπει να έχουν χώρο ύπαρξης και γι' αυτό πιστεύουμε ότι το 7% στην πρόταση της Κομισιόν είναι θετικό βήμα πρόοδου. Μπορεί σε μερικά χρόνια να διαπιστώσουμε ότι χρειάζεται ε, να αυξηθεί το ποσοστό σε 10-15%. Αλλά κυρίως ε, στις ε, περιοχές εντατικής γεωργίας θα πρέπει να διατηρήσουμε ή να ξαναδημιουργήσουμε διαδρόμους οικολογικούς να αποκαταστήσουμε ε, κάποια περιβάλλοντα. Είναι ε, ζωτική σημασία να διατηρήσουμε αυτούς τους διαδρόμους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Αντιπρόεδρε Πόλσον, ο Άλμπερτ Τες και μετά η Μαρία Νεντελτσέβα. Χωρίς μικρόφωνο, ο κύριος oh. Und BDA konnte nicht pünktlich hier sein, deshalb Ζήτω συγγνώμη που δεν... Ο Πετεριά δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ στην ώρα του, γι' αυτό πρώτα θα παρουσιάσω τις δικές του θέσεις και κατόπιν θα υποβάλω τα δικά μου σχόλια. Ε, ε, γενικά μπορούμε να επικροτήσουμε την ε, θέση της κυρίας. θα πρέπει να διατηρηθεί η βιοπικιλότητα και θα πρέπει να ληφθούν απαραίτητα μέτρα. Επιπλέον θα πρέπει να... Ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πετύχει βελτιώσεις στον τομέα της βιοπικιλότητας. Και οι προτάσεις ε, της Κομισιόν ε, είναι πολύ θετικές και θα πρέπει να αυξηθεί ε, στο 10% ε, το ποσοστό των ε, οικολογικών περιοχών και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις σχετικές οδηγίες όπως αυτές για τα ύδατα και, την, την, και τα προϊόντα φυτοπροστασίας. Οι δικές μου παρατηρήσεις είναι οι εξής. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά σε αντικειμενικό επίπεδο, διότι θα πρέπει να είναι σαφές το εξής. Όταν ε, προστατεύουμε περιοχές, πρόκειται για περιοχές οι οποίες ε, φτάσανε στην κατάσταση που βρίσκονται επειδή δεν ε, είχαν προστατευτεί. Γιατί χρειάζεται να προστατεύσουμε περιοχές οι οποίες χωρίς προστασία μέχρι στιγμής έχουν συμβάλει στη βιοπικιλότητα έχει υποθεί ότι όσο η πολιτική και η διαχείριση δεν ε, υπαγόρευε τίποτα στους ε, αλείς και στους ε, κυνηγούς προστάτευαν τις αντίστοιχες περιοχές αλλά όταν επιβλήθηκαν μέτρα οι ε, δεν συνέβαλαν σημαντικά στην βιοποικιλότητα, διότι ένιωθαν ότι ότι τους πίεζαν πολύ τα μέτρα αυτά και το θέμα είναι μήπως ε, χωρίς προστασία έχουν λειτουργήσει καλύτερα οι περιοχές αυτές. Δεν θα είχα αντίρρηση εάν κάποιες ε, αστικές ε, περιοχές προστατεύονταν. Στην Γερμανία έχει γίνει μια έρευνα και διαπιστώθηκε ότι την μεγαλύτερη βιοπικιλότητα έχουν κάποια προάστια πόλεων. Μήπως ε, θα έπρεπε τέτοιες περιοχές να προστατευτούν οικολογικά επιπλέον. Όσον αφορά την ε, βιοπικιλότητα υπάρχουν εδώ σημαντικές αντιφάσεις. Επί 12 χρόνια ε, ασχολούμουν με θέματα τέτοιας διαχείρισης. Στην χώρα μου έχει χτιστεί το κανάλι του Δούναβη ε, τώρα όταν ε, ένας ε, εργολάβος θέλει άδεια για λατομείο δεν δίδεται η άδεια διότι αυτό εμποδίζει την βιοπικιλότητα. Έχουμε όμως ένα λατομείο το οποίο δεν μπορούν να το ξαναγεμίσουν διότι έτσι θα καταστραφεί η βιοπικιλότητα. Τώρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να αλλάξει τίποτα λόγω της βιοπικιλότητας. Κάτι παρόμοιο συνέβη στην περιοχή μου. 100 ε, ε, ε, εκτάρια είχαν οι Αμερικάνοι για είχαν ε, εκεί μια περιοχή, αλλά αν θα ήθελε σήμερα κανείς να δημιουργήσει μια τέτοια περιοχή, ε, δεν θα ε, επιτρεπόταν. Ωστόσο, σε αυτήν την περιοχή υπάρχει σήμερα η μεγαλύτερη βιοπικιλότητα. Και ένα τρίτο παράδειγμα έχω ακόμα να σας δώσω, τη δεκαετία του 1960 έγινε αποξήρανση μια, ενός ε, υδροβιότοπου. Ε, σήμερα δεν θα επιτρεπόταν κάτι τέτοιο. Ε, σήμερα όμως υποτίθεται ότι αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για, για γεωργική έκταση. τώρα ε, καλλιεργούνται τα εδάφια αυτά, ωστόσο θεωρείται ότι θα πρέπει να προστατευτούν ε, εκεί κάποια πουλιά που έχουν κατασταθεί εκεί. Ε, μήπως θα πρέπει να διδάξουμε τα πουλιά να μην πηγαίνουν εκεί επειδή δεν, ε, συνάδουν, ε, δεν ε, ακολουθούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να βρούμε το σωστό τρόπο, διότι θέλουμε να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα, δεν θα πρέπει όμως απλά να στυλιτεύουμε τη γεωργία, διότι η γεωργία και στην Ευρώπη συμβάλλει σημαντικά στην προστασία της βιοπικιλότητας και δεν θα πρέπει να τους παρενοχλούμε τους γεωργούς θα πρέπει να του δώσουμε κίνητρα ώστε να, διατη... να βοηθάνε και αυτή τη διατήρηση τη βιοπικιλότητα. Μάλιστα, ευχαριστούμε Άλμπερτ και τώρα έχει το λόγο η Μαρία Νεντελτσέβα και μετά ο κύριος Φεϊμό. Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εισήγησή της που είναι εξαιρετικά χρήσιμη και να συνδέσω τα μέτρα που προτείνει η συγγήτρια όσον αφορά τη βιοπικιλότητα με την νέα κοινή γεωργική πολιτική που είναι πιο οικολογική και πιο πράσινη. Θα ήθελα να ασχοληθώ με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τομείς που προωθούν τη βιοπικιλότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι η μελισσοκομεία είναι ένα τέτοιο τομέα. Οι μελισσοκόμοι αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή μεγάλα προβλήματα. Όμως ο τομέας αυτός είναι πολύ σημαντικός για την επικονίαση και κατά συνέπεια για την ε, βιολογική ποικιλία, πολυμορφία. Η νέα η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να λάβει υπόψη όλους τους στόχους που περιλαμβάνονται σε αυτή την πρόταση και οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε όλα τα μέτρα που προτείνονται είτε να μπορέσουν να ενταχθούν μέσα στην κοινή γεωργική πολιτική. Πρέπει δηλαδή να προωθήσουμε και να βοηθήσουμε τους μελισσοκόμους ώστε να υλοποιήσουν τους στόχους τους, καθώς μάλιστα μιλάμε για νέα πράσινα μέτρα θα μπορούσαμε να, τους, να προβλέψουμε κάποια βοήθεια, να βρούμε μέσα ώστε να τους παροτρύνουμε να επενδύσουν στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι για τις προτάσεις σας. Ευχαριστούμε Μαρία. Το λόγο έχει ο κύριος Φαϊμόν και μετά η κυρία Κλάς. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπε ο συνάδελφος Άλμπερτ Ντες. Εγώ μένω κοντά σε μια παλιά σοβιετική στρατιωτική βάση. Σύμφωνα με τους δικολόγους μας ε, ανακάλυψαν ότι αυτή η στρατιωτική βάση ήταν και ζώνη βολής και είναι ταυτόχρονα μια ζώνη μεγάλης βιοπικιλότητας. Γι' αυτό τον λόγο σε αυτή την περιοχή βολής είχε απαγορευτεί η γεωργία και κάποιες φορές υπάρχει η βιοπικιλότητα σε μέρη όπου δεν θα το περίμενε κανείς. Αυτή ήταν μια παρατήρηση σχετική με το θέμα. Η δεύτερη μου παρατήρηση αφορά τις προσπάθειες για διεύρυνση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εγώ έρχομαι συχνά σε επαφή με γεωργούς και τους μιλώ για τα μέτρα που προετοιμάζουμε στις Βρυξέλλες και πάντοτε στο τέλος μου θέτουν την εξή ερώτηση. Πιστεύετε ότι εσείς στην Βρυξέλλες γνωρίζετε καλύτερα από ότι ένας χωρικός που ζει εδώ, ένας αγρότης που ζει εδώ επί τόπου, μέσα στη φύση, στο αγρόκτημά του για πολλές γενναίες νομίζετε ότι ξέρετε καλύτερα τι πρέπει να γίνει εδώ. Πιστεύετε πως καλύτερα θα τα σχεδιάσετε από τις Βρυξέλλες το τι πρέπει να κάνουμε εμείς, εμείς που διαχειριζόμαστε αυτή την περιοχή εδώ και γενιές και σας ομολογώ ότι συχνά δεν ξέρω τι να απαντήσω. Είναι περίπλοκο το θέμα και εν γέννη, εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον της βιοποικιλότητας, αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε και τι θα σημάνει αυτό ως απέτηση σε σχέση με τους γεωργούς. Αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να φτιάξουμε μέτρα απλά, τα οποία δεν θα επιβαρύνουν τη γραφειοκρατία για τους ε, γεωργούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φάιμον. Η κυρία Κλάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η βιοπικιλότητα μου φαίνεται πως είναι σύνθημα. Το συζητά, τη, συζητάμε σε ε, πολλές επιτροπές και ο καθένας έχει δικές του ιδέες ε, στο μυαλό του και ο καθένας ε, ε, ερμηνεύει διαφορετικά τη λέξη αυτή και επιδιώκει να πετύχει τα δικά του συμφέροντα. Εμείς τι θέλουμε, βιοπικιλότητα σημαίνει διατήρηση. Ε, εάν ναι, τότε δεν αρκεί να μην κάνουμε τίποτα. σήμερα ήρθα από μια συνέλευση στην εκλογική μου περιφέρεια. μου είπαν ότι ε, έχουν πρόβλημα στις ε, φοιτίες τους ε, λόγω ενός φυτού το οποίο προστατεύστηκε πριν μερικά χρόνια διότι επειδή ήταν ένα είδο ε, υποαπειλή πριν κάποια χρόνια, τώρα όμως ε, δημιουργεί υπερβολικά πολλά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν τα μέτρα να ληφθούν την κατάλληλη στιγμή. Ε, η διατήρηση δεν μπορεί να γίνει εάν δεν λάβουμε υπόψη μας και την γεωργία. Στην έκθεση θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο 2. Δεν μπορούμε εδώ να προδικάσουμε άλλες αποφάσεις. Θα πρέπει η βιοπικιλότητα να είναι θέμα των περιφερειών, οι περιφέρειες οι ίδιες ε, να ε, το ρυθμίζουν αυτό και να λαμβάνουν μέτρα όπου είναι απαραίτητα και σημαντικά. Ευχαριστώ. Bene, adesso, eh, la parola. Sì. Μάλιστα, τώρα ο Μισελ, ο Μισελ Νταντέν ζήτησε το λόγο και μετά θα πάρει το λόγο η Κομισιόν. Κύριε Πρόεδρε, για αυτό το θέμα της βιοπικιλότητας, πιστεύω πως όντως από την μια περιοχή στην άλλη, τα αποτελέσματα μπορούν να διαφέρουν σε σχέση με τις πρακτικές. Ε, μέχρι στιγμής, στο δεύτερο πυλώνα, ε, προσανατολιστήκαμε κυρίως σε μέτρα που απαιτούν ε, πόρους περισσότερο από ό,τι σε μέτρα που στόχο έχουν να αποζημιώσουν το αποτέλεσμα. Και για αυτό το θέμα της βιοπικιλότητας πιστεύω πως η Επιτροπή μας θα έπρεπε να επιμείνει για την ανάγκη επίτευξη αποτελεσμάτων. Και όταν μιλάμε για αποτελέσματα σημαίνει ότι θα αφήσουμε τον Γιωργό να κάνει ό,τι νομίζει γιατί γνωρίζει την περιοχή του στα εθνικά Πάρκα ξεκίνησε ένα μέτρο μέσω που ονομάζεται Ανθισμένα Πάρκα, ένα μέτρο που, στο οποίο συμμετέχουν οι Γεωργοί και ε, που είναι πολύ επιτυχές, ενώ προηγούμενα στις ίδιε περιοχέ είχαμε προσπαθήσει να φτιάξουμε υποχρεωτικά μέτρα που όμως αυτά δεν έδωσαν αποτελέσματα. Επίσης, συχνά μιλάμε εδώ για το θέμα της μελισσοκομείας. Πρόσφατα είδα αποτελέσματα για το μίσο που μια διαφοροποίηση των καλλιεργιών και κυρίως ε, η χειμερινή κάλυψη των, καλλιεργιών ε, είχε προβλεφθεί και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά και για την μεθεπόμενη χρονιά παραγωγής μελιού. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ε, Μισελ, και τώρα το λόγο θα πάρει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο Διευθυντής Βάκενχουτ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την πλούσια συζήτηση που έγινε απόψε για αυτή την ε, ουσιαστική διάσταση του μέλλον, για το μέλλον της βιοπικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ, πολλές από τις παρεμβάσεις τόνισαν ιδιαίτερα την ευθύνη της γεωργίας και τον ανάγκη, την ανάγκη να αντιμετωπιστούν και άλλοι τομείς ταυτόχρονα. Μπορώ να σας καθησυχάσω, είναι σαφές πως η, βιοπικιλότητα σημαίνει ευθύνη όχι μόνο γιατί η γεωργία και η δασοκομεία καλύπτουν το 72% της επικράτειας της Ένωσης, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να αναζητήσουμε αλλού τομείς σε άλλου τομεί τι θέλουμε να κάνουμε. Και αυτό ακριβώς κάνουμε με αυτή την στρατηγική της βιοπικιλότητας. Έχουμε περιγράψει έξι στόχους. Ο ένας ε, εστιάζει στη γεωργία και έχει έναν ε, ε, μικρότερο στόχο για τη δασοκομεία και οι άλλοι εστιάζουν σε άλλους τομείς μεταξύ των οποίων και η αλληλεία που αναφέρθηκε από κάποιους από εσά, αλλά και η γενική πράσινη υποδομή όπως αποκαλείται που συνδέεται με συστήματα οικοσυστημάτων με, με υπηρεσίες οικοσυστημάτων, με συγχωρείτε. Όσον αφορά συνολικά την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, θα πρέπει να τονίσουμε, όπως έγινε από διάφορους ομιλητές, πως ήδη έχουν επιτευχθεί πολλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο χάρη στους πόρους που δόθηκαν μέσω των ευρωπαϊκών διόδων για μέτρα στήριξη στην Ένωση, καθώς και τα πολύ καλά αποτελέσματα για τη βιοπικιλότητα από ορισμένε πτυχές της γεωργικής μας πολιτικής. Πρέπει ωστόσο να αναγνωρίσουμε πως και άλλα πρέπει να γίνουν και γι' αυτά έχουμε στοιχεία και αυτά τα στοιχεία φυσικά έχουν ε, χρησιμοποιηθεί Είναι όμως κάποια στοιχεία προβληματικά όσον αφορούμε την κατάσταση των ειδών που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Βλέπουμε τότε πως δεν βρισκόμαστε ακόμα εκεί που θα θέλαμε. Το 17% αυτών των ειδών είναι σε καλή κατάσταση ε, διατήρησης, αλλά δεν είναι αυτό ικανοποιητικό και στις γεωργικές περιοχές αυτό το ποσοστό είναι χαμηλότερο. Και αυτό φυσικά σημαίνει περισσότερη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποια στοιχεία που νομίζω είναι σημαντικό να τα ξανα να αναφέρουμε είναι η σύνδεση ανάμεσα στην ε, διατήρηση και τη βιώσιμη παραγωγή. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την διατήρηση, τη συντήρηση, γιατί ορισμένες παρεμβάσεις ανέφεραν ήδη πως στο παρελθόν, την παρελθούσα δεκαετία εκεί ήμασταν πολύ δραστήριοι. Όντως εδώ έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο 18% σε σχέση με το ποσοστό ε, της ευρωπαϊκές επικράτειες που αντιπροσωπεύουν και που είναι προστατευόμενες. Πολλές από αυτές τις περιοχές βρίσκονται σε γεωργικές περιοχές και ε, συνορεύουν με γεωργική γη. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε είναι τι γίνεται με το υπόλοιπο 82% ε, που δεν προστατεύεται. Βιώσιμο τρόπο δηλαδή παραγωγής που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της παραγωγής τροφίμων αλλά δεν θα υποβαθμίζει τη βιοπικιλότητα στην Ένωση. Και ως προς αυτό, οι προτάσεις που έχουμε θέσει, που έχουμε υποβάλει, δίνουν τέτοια ισορροπία. Δεν υποχρεώνουν, αλλά ε, οδηγούν, παροτρύνουν για συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους τομείς, γεωργία και δασοκομεία, γιατί αυτό που είναι σαφές είναι ότι δεν θα επιτύχουμε τους στόχους βιοποικιλότητας χωρίς την ισχυρή και συνεχή εμπλοκή του τομέα, που ούτως ή άλλως ήταν ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους σε όσα προσπαθήσαμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ. Molto Ωραία, ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις σας και τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Ντάντσιλα για να ακούσουμε τα δικά της σχόλια και μετά να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όλες τις προτάσεις των συναδέλφων καθώς και τα προβλήματα τα οποία έχουν ε, θυγεί. Νομίζω ότι ε, επανειλημμένως άκουσα δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα πόσο σημαντική είναι η βιοπικιλότητα και επίσης πολλοί συνάδελφοι εξέφρασαν ε, την ανησυχία μήπως επιβαρύνει η διατήρηση τη βιοπικιλότητα πολύ περισσότερο τους ε, αγρότες. Ε, μιλήσατε για το Δούναβι, κύριε Ντές, ε, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμο στην ιδιαίτερη σα πατρίδα. Αλλά θα πρέπει να σα πω ότι η κατάσταση με το Δέλτα του Δουνάβεω είναι τελείω διαφορετική στην περιοχή του κυρίου Ντε. Από εκεί μάλλον υπάρχουν πολλά προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε εξαφάνιση πολλών ειδών. Και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε κάποιες κοινέ λύσεις που θα μπορούν να ε, ικανοποιήσουν ε, τις ανάγκες όλες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε ό,τι αφορά το επίπεδο προστασίας της βιοπικιλότητας. Πιστεύω επίσης ότι αυτό το θέμα πρέπει να τύχει μεγαλύτερης προσοχής και ίσως θα ήταν καλό να είχαμε και περισσότερο χώρο, να είμαστε είχαμε μια πιο μακροσκελή γνωμοδότηση, αλλά ξέρετε ότι είναι περιορισμένη η έκταση μιας γνωμοδότησης. Πάντως ο στόχος μου είναι να είμαι ω δυνατόν πιο πλήρης σε αυτή την γνωμοδότηση και να επικεντρωθώ στα πραγματικά προβλήματα που αφορούν και την βιοπικιλότητα και την Ευρωπαϊκή Γεωργία συγχρόνως. Ωραία, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συζήτηση. Να σας θυμίσω ότι η παρουσίαση, των βολήμαλων τροπολογιών, έχει οριστεί για τις 7 Φεβρουαρίου στις 12. Λιγότερα από μία μέρα έχουμε προθεσμία δηλαδή. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερής της διάταξης και με τη συζήτησή μας στρεφόμαστε στη μεταρρύθμιση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής που φυσικά θα είναι η προτεραιότητα για φέτος. <coughs> Μετά από τη συζήτηση που έγινε στην τελευταία μας συνεδρίαση, όπου όπως θα θυμάστε συζητήσαμε για άμεσες πληρωμές και για ενιαία κόα, τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε πιο ενδελεχώς τις προτάσεις της Κομισιόν για την ανάπτυξη της υπαίθρου και για τον οριζόντιο κανονισμό για τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ. Οι δυο μας εισηγητές, ο Λουίς Μανουέλ Καπούλα Σάντος και ο Τζοβάνι Λαβία, είναι εδώ. Το Λουίς τον βλέπω. Ο Τζοβάνι Λαβία που να είναι καταφθάνει, πιστεύω. Credo sia importante, cari colleghi, ricordare... Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω πως είναι σημαντικό να θυμόμαστε την ανάγκη ύπαρξης ισορροπίας ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ. Είναι σημαντικά τα προγράμματα για να διατηρηθεί η πολυμορφία των περιοχών της υπαίθρου στην Ευρώπη και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν και έτσι με μεγάλη μου χαρά δίνω το λόγο στο Λουίς για να ανοίξει αμέσως τη συζήτηση για την νομοθετική πρόταση για την ανάπτυξη υπαίθρου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι. Μπαίνουμε στην καθοριστική φάση της διαδικασίας μεταρρύθμισης και πρόκειται για έναν κανονισμό πολύ σημαντικό. Είναι ένας πολύ σημαντικός κανονισμός που δεν μπορεί να συζητηθεί χωριστά από τον κανονισμό περί άμεσων πληρωμών. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι ένα σύνολο, αποτελείται από δύο πυλώνες και το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι θα έπρεπε να έχει δύο πυλώνες η δημοσιονομική κατανομή κατά βάση διαφέρει, ε, μάλλον διαφέρει πολύ σημαντικά από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Η λογική εφαρμογή φυσικά είναι πολύ διαφορετική, όμω είναι δύο πραγματικότητε αδιαχώριστε και δεν μπορεί κανεί να δει την κοινή γεωργική πολιτική βλέποντα μόνο τον ένα πυλώνα. Θα ήταν σαν να κοιτά έναν άνθρωπο και να βλέπει μόνο και να, κοιτώντας, να κοιτάς έναν άνθρωπο και να βλέπεις μόνο τον μισό. Έχουμε λοιπόν έναν μεγάλο κατάλογο μέτρων που μας προτείνει η Κομισιόν, πάνω από δύο δεκάδες. Είναι δύσκολο να μην συμφωνήσουμε με, τις περισσότερες από αυτές, γιατί, με τα περισσότερα από αυτά, γιατί είναι θετικά μέτρα που έχουν προετοιμαστεί καλά και που αξίζουν την στήριξή μας. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες πτυχές που πρέπει να διορθώσουμε, να διευκρινίσουμε και να βελτιώσουμε. Όμως η Κομισιόν σε αυτή τη διαδικασία έχει οθετήσει μια συμπεριφορά πολύ διαφορετική από την προσέγγιση που έκανε ε, στην πρώτο πυλώνα από αυτή με το δεύτερο πυλώνα. Γιατί στο πρώτο πυλώνα μας κάνει μια πολύ αντικειμενική πρόταση κατανομής των δημοσιονομικών πόρων ανακράτους μέλος. Στο δεύτερο όμως πυλώνα η Κομισιόν έχει παραλείψει αυτό το θέμα και μας ζητά να της δώσουμε μια λευκή επιταγή, ώστε η Κομισιόν να κάνει τη δημοσιονομική κατανομή που θεωρεί κατάλληλη, χρησιμοποιώντας δύο στόχους μόλις. Ο ένας είναι ότι τα προγράμματα κάθε ενός από τα κράτη-μέλη θα σέβεται τους τρεις ε, στόχους, το πράγμα που θεωρώ εύκολο να στηρίξουμε, και έπειτα το δεύτερο κριτήριο είναι τα προηγούμενα αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτή η φράση. Σημαίνει ότι γίνεται μια αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εγώ δεν ε, συμφωνώ όμως ότι εμείς στο Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της συναπόφασης, να καθόμαστε να συζητάμε την ε, κοινή γεωργική πολιτική και να μπορούμε μόνο να συζητάμε ένα κομμάτι της, του προπολογισμού της, ακόμα και αν είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, γιατί η δεύτερη πρόταση της Κομισιόν, όπως ξέρετε, το 65% είναι στο πρώτο πυλώνα και 25% είναι ε, στον δεύτερο πυλώνα και τα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται σε καλύτερη θέση ε, στον πρώτο πυλώνα βρίσκονται σε χειρότερη θέση στο δεύτερο πυλώνα και τούμπαλιν. Και κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να έχουμε μια σοβαρή προσέγγιση στην κοινή γερική πολιτική και τη μεταρρύθμισή της αν δεν εξετάσουμε τους δύο πυλώνες μαζί. Και γι' αυτό και σκοπεύω να κάνω μία πρόταση μέσω της δικής μου έκθεσης, να λάβω αυτή την πρωτοβουλία δηλαδή, μία πρόταση προϋπολογισμού για το δεύτερο πυλώνα, με βάση τα όσα έκανε η Κομισιόν στον πρώτο πυλώνα και θα προσπαθήσω στην έκθεσή μου να παρουσιάσω μια συσχέτιση ανάμεσα στην ε, δημοσιονομική πρόταση του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για σύγκληση στους δύο πυλώνες από κοινού και όχι μόνο στα ένα. Γιατί δεν έχει νόημα να μιλάμε για σύγκληση στα κράτη-μέλη μόνο για τον πρώτο πυλώνα και να αφήσουμε ε, τα υπόλοιπα στο δεύτερο πυλώνα όπω είναι. Ή να περάσουμε σε μια μεταρρύθμιση την οποία θα κάνει από μόνη τη η Κομισιόν όπως νομίζει, όπω κρίνει. Είναι πολύ ευαίσθητη αυτή η πολιτική και πρέπει να αποφασίσουμε την πολιτική μα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιε είναι οι δικές σας ε, απόψεις σχέση με αυτή την προσέγγιση. Σας λέω ποιες είναι οι επιλογές. Να στηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν και να αφήσουμε την Κομισιόν να αποφασίσει ό,τι νομίζει ή το Κοινοβούλιο να λάβει μια πρωτοβουλία και να υποβάλει δική του πρόταση και να την εντάξει στο ευρύτερο πλαίσιο της ανακατανομής των πόρων ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στους ε, γεωργούς. Πέρα από αυτό, άλλα λεπτά ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε είναι το θέμα των ε, λιγότερο ευνοημένων περιοχών. Εδώ η Κομισιόν προτείνει ότι τα κράτη-μέλη να προτείνουν ε, την προοπτική περιορισμού. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να εγκρίνουμε πάλι ως Κοινοβούλιο μια ειδική παρέμβαση χωρίς να ξέρουμε ποια είναι αυτή η ειδική παρέμβαση, ανεξάρτητα δηλαδή από τους όρους που θέτει η Κομισιόν για να είναι επιλέξιμη η στήριξη. Κάτι ακόμα που πρέπει να αποσαφινιστεί είναι το θέμα της διαχείρισης κινδύνων και πιο συγκεκριμένα ο μηχανισμός σταθεροποίησης των ε, αποδοχών. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς το μηχανισμό που προτείνει η Κομισιόν γιατί εντάξει εγώ το καταλαβαίνω αλλά λέει η Κομισιόν ότι για τα ε, ταμεία κεφαλαίων, τα αρχικά, δεν είναι δυνατόν να γίνει δημόσια επένδυση. Αυτό σημαίνει πως η γεωργοί θα πρέπει οι ίδιοι να χρηματοδοτήσουν το αρχικό κεφάλαιο των ε, συνεταιρισμών τους θα λειτουργήσουν με αυτό το αρχικό κεφάλαιο και με δάνεια και μόλις θα υπάρξει συμμετοχή δημόσια, αφού θα έχει αρχίσει δηλαδή να λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Νομίζω πως είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε αυτή την κατάσταση που γνωρίζουμε ότι ισχύει σε πάρα πολλές περιοχές πολλών κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να διευκρινιστεί. Γιατί Αυτός ο μηχανισμός δεν έχει καμία πρακτική αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιό να μας εξηγήσει κάπως καλύτερα σήμερα εδώ για όλους μας να μας εξηγήσει ποιος ακριβώς είναι ο μηχανισμός χρηματοδότησης που προτείνει και συγκεκριμένα για το μέσο σταθεροποίησης των εισοδημάτων. Επίση, η Κομισιόν προτείνει μια, ένα αποθεματικό αποτελεσματικότητα. Αυτό σημαίνει πω τα κράτη-μέλη που έχουν πιο καλούς διοικητικού μηχανισμούς θα έχουν πλεονεκτήματα σε σχέση με τα πιο μικρά κράτη που έχουν λιγότερο αποτελεσματικούς διοικητικού μηχανισμούς και νομίζω πως ε, να υπάρχει ένα δημοσιονομικό απόθεμα για αυτούς που ήδη βρίσκονται σε καλύτερη θέση δεν είναι πολύ λογικό. Επίσης γίνεται λόγος για 25% του φακέλου για την ε, γεωργική ανάπτυξη για τα περιβαλλοντικά μέτρα. Και πάλι δεν γίνεται λόγος για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το μόνο συγκεκριμένο πράγμα είναι το 5% για το leader. Θέλω να ακούσω τη γνώμη των συναδέλφων λοιπόν και με βάση τη γνώμη σας να προσπαθήσω να συντάξω μια έκθεση που να αντιστοιχεί στις προσδοκίες των περισσότερων έξιμων. Αλλά όπως σας είπα το πρώτο θέμα επί το οποίο θα πρέπει να λάβουμε απόφαση στις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες αφορά το θέμα της χρηματοδότησης και οι επιλογές είναι δύο. Είτε δεχόμαστε ότι η Κομισιόν θα αποφασίζει χωρίς το Κοινοβούλιο να έχει λόγο ή να τολμήσουμε να προτείνουμε εμείς μια πρόταση δημοσιονομική, γνωρίζοντας ποιες είναι οι δυσκολίες και τις αντιφάσεις που σίγουρα θα υπάρχουν μεταξύ μας. Πάντως, πρόθεσή μου είναι να κάνω μια πρόταση προϋπολογισμού και να τη συνδέσω με την δημοσιονομική πρόταση του πρώτου πυλώνα, ώστε να υπάρξει μια σφαιρική προσέγγιση του προϋπολογισμού της κοινή γεωργικής πολιτικής και του προβλήματος της ανακατανομής. Έχω και άλλα πολλά να πω, Πρόεδρε, αλλά δεν θέλω να μονοπολίσω τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε περαιτέρω. Ε, Ευχαριστώ, Λουίς. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτος ο κύριος Καλινόσκη και, μετά η Αντιπρόεδρος Πόλσον. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω να διατυπώσω αρκετές παρατηρήσεις. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ σε δύο τουλάχιστον και μετά να κάνω και μια ερώτηση. Το σχέδιο κανονισμού φαίνεται να βάζει πολύ μεγάλη έμφαση στο δεύτερο πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική οικονομία στην Ήπεθρο και επικεντρωνόμαστε και στις νέες προκλήσεις. Σίγουρα δεν χωρεί αμφιβολία στο ότι υπάρχει ανάγκη να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Να προστατεύσουμε επίσης και το κλίμα μέσω της προστασίας της βιοπικιλότητας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε επίσης νέα δίκτυα. Όλα αυτά τα θέματα όμως δεν θα πρέπει να αποτελέσουν ε, τη μόνη μας, ε, το μόνο μας επίκεντρο. Έχουμε τους στόχους ε, στο δεύτερο πυλώνα, αλλά τι γίνεται με τη μεταποιητική βιομηχανία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν ε, και διορθωτικά προβλήματα. Δεν βλέπω να γίνεται κάποια αναφορά σε αυτά. Και έρχομαι στο δεύτερο σχόλιο. Αρχή επικουρικότητας και πού θα βασιστεί ο προγραμματισμός. Ανάλυση των αναγκών. Όλα αυτά ε, με δημιουργούν κάποιες ανησυχίες ό,τι αφορά τον κανονισμό. Δεν νομίζω ότι ρυθμίζονται με το σωστό τρόπο, γιατί παραμένει η ευθύνη στα κράτη-μέλη ή μήπως θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία τα κράτη-μέλη στη διάθεσή τους. δεν νομίζω ότι θα έχουμε να αποκομίσουμε κάτι θετικό. Με αυτά τα ποσά το οποία διατίθεται 5% για το Leader και 25% για τα άλλα προγράμματα. Και αν μου επιτρέπετε ένα ερώτημα. Η Οργανισμοί πληρωμών, μήπως θα πρέπει να επαναπιστοποιηθούν για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Αντιπρόεδρος Πόλσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, διότι ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Σάντος. Υπάρχουν πάρα, πάρα πολλές λεπτομέρειες στο πρόγραμμα για την Ήπεθρο και με τρομάζει αυτό λίγο, διότι κάθε μικρό πρόγραμμα ακολουθείται από ε, ε, ανακοίνωση ότι θα ακολουθήσει μια πράξη κατοξιδότηση και τελικά θα καταλήξουμε σε ιδιαίτερα πολύπλοκη νομοθεσία. Θα ήθελα όμως επίσης να σας καλέσω να κοιτάξουμε λίγο όλη την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Περνάμε οικονομική κρίση, περνάμε τραπεζική κρίση. Έχουμε αυξημένη ανεργία και έχουμε μία ύπεθρο που εγκαταλείπεται από τον κόσμο. Ακόμα και στη δική μου χώρα που ανήκει στις τρεις ή τέσσερις ε, χώρες της Ένωσης ε, που σε κρατικό επίπεδο έχει πολύ καλή οικονομία. Ε, ακόμα και στη χώρα μου λοιπόν έχουμε ανεργία των νέων ε, που φτάνει τα 20% ιδιαίτερα στην Ήπεθρο. Έχουμε Ήπεθρο που, που φτωχαίνει ε, με ραγδαία ταχύτητα. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου τις εικόνες αυτές όταν συζητάμε τις λεπτομέρειες του προγράμματος για την Ήπεθρο και θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς μπορεί το πρόγραμμα αυτό να αποτελέσει εργαλείο σε αυτό το συνολικό παιχνίδι, διότι η Ευρώπη και κυρίως η Ήπεθρός μας δεν μπορεί να περάσει την κρίση αυτή με περικοπές. Δεν αρκεί να περικόψουμε τους προϋπολογισμούς, θα πρέπει να φροντίσουμε κάθε ευρώ να χρησιμοποιείται σωστά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Και θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποιες λεπτομέρειες. Καταρχήν, θα ήθελα να ε, ασχοληθούμε με τον κανονισμό ομπρέλα όπου εμπίπτει ε, η πολιτική αλληλείας, ε, η πολιτική πέθρου και η αγροτική πολιτική. Θα μπορέσουμε εκεί να βρούμε χρηματοοικονομικούς ε, πόρους ώστε οι αγρότες και οι άλλοι παράγοντες να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια κινδύνου. Δεν θα έχουν τέτοια πρόσβαση τα επόμενα χρόνια εάν κοιτάξουμε την ε, πραγματικότητα στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Υπάρχει εδώ δυνατότητα για δημιουργία, για καινοτομία, για ελευθερία και ίδια ευθύνη για τους ενθουσιώδεις ανθρώπους ε, στην ε, Ήπεθρο, διότι έχουμε πολύ ικανούς ανθρώπους αρκεί να τους στηρίξουμε. Άλλες ε, δύο λεπτομέρειες ε, στις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ ε, είναι καταρχήν το θέμα των ζώων. Στον τομέα 1 μιλάμε για εκτάσεις και χρήματα. Στον πυλώνα 2 ασχολούμαστε με τις λεπτομέρειες. Αυτό είναι σαφές. Νομίζω ότι η προστασία των ζώων ανήκει στα θέματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αποτελεί αυτό σημαντικό παράγοντα και για, τον, για την ανάπτυξη και για το περιβάλλον και για την καινοτομία. Η γεωργία και η δασοκομεία θα πρέπει να είναι αυτάρκης όσον αφορά την ε, ενέργεια και εννοώ να χρησιμοποιούνται τα απόβλητα για την παραγωγή ενέργειας, όχι να υπάρχει παραγωγή ενέργειας στις γεωργικές εκτάσεις. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους σπόρους ώστε να πετύχουμε βελτίωση για ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Αντιπρόεδρο Πόλσον και τώρα θα δώσω το λόγο στον Τζαν Σκοτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας ένα συγκεκριμένο και πολύ σημαντικό ζήτημα που είχα αναφέρει και τον Οκτώβριο όταν είχα υποβάλει σχετική προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν. Μιλώ συγκεκριμένα για τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ταμείου εγγύησεων που θα παρέχει δάνεια σε νέους αγρότες, σε νεαρούς αγρότες. Το άρθρο 18 του σχεδίου κανονισμού, σε ό,τι αφορά το Γεωργικό Ταμείο, ήδη κάνει λόγο για στήριξη και των υλικών και των άλλων επενδύσεων. Και σε ό,τι αφορά τα μέγιστα ποσά, τα οποία αναφέρονται, ε, δεν είναι και τόσο υψηλά, αλλά αν έχουμε μία ε, προσάξη κατά 20% για τους νεαρούς εργότες θα ήταν ε, καλύτερο. Ένα άλλο άρθρο το οποίο μιλά πάλι για την παροχή βοήθεια στους νεαρούς αγρότες, μιλά πάλι για ένα μέγιστο ποσό. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου αυτού ορίζεται το σχετικό ποσό οι δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να ζητήσουν από τους αρμόδιους οργανισμούς πληρωμών μια προκαταβολή η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των δημόσιων ενισχύσεων σε επενδύσει. Η απάντηση της Κομισιόν στην προφορική ερώτηση που είχα υποβάλει ήταν θετική. Έλεγε δηλαδή ότι στο πλαίσιο του κοινού στρατηγικού πλαισίου για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ενδεχομένω θα μπορούσαν να διατεθούν ε, ταμεία εγγύησεων αλλά και κάποια κεφάλαια για δανεισμό για τους νέους ε, αγρότες. Πρέπει νομίζω να μιλήσουμε συγκεκριμένα για αυτό το ταμείο. Ναι, μεν προβλέπονται και ενισχύσεις ε, και επιδοτήσεις. Ένα τέτοιο ταμείο θα έδινε περισσότερα κίνητρα στους νεαρούς αγρότες για να εργαστούν ε, στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η Ερνάνθ ε, Γκαρσία τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Καπούλας γιατί συζητούμε με τις προτάσεις του αυτό το σκέλος ε, της της πολιτικής. Η πρόταση μας δημιουργεί κάποια προβλήματα η Ισπανία, όπως ξέρετε, είναι μια χώρα που έχει ένα ε, σύστημα γεωργικών ασφαλίσεων κρατικών και θα μπορούσε έτσι να προκύψει πρόβλημα με τη συμβατότητα ή μη συμβατότητα του ήδη φυστάμενου στην Ισπανία συστήματος. Και θα ήταν κρίμα μια προσπάθεια βελτίωσης των ε, πραγμάτων και της κατάστασης ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιδεινώσει την κατάσταση σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Επομένως η αντιπροσωπεία μου πραγματικά θα δώσει πολύ μεγάλη προσοχή στο να ε, διασφαλιστεί η συμβατότητα ε, του συστήματο που έχει δρομολογηθεί και ισχύει εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μου την Ισπανία με αυτά τα οποία προτείνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα επίση να αναφέρω ένα πρόβλημα το οποίο εμεί ω Ισπανία αντιμετωπίζουμε. Γνωρίζετε ότι η Ισπανία είναι η πλέον αποκεντρωμένη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τι αυτονομίε Έχουμε δηλαδή μεταφορά αρμοδιοτήτων, εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το Ισπανικό κράτος ε, στις αυτόνομε περιφέρειες. Και έτσι έχουμε 16 σχέδια ανάπτυξης τη υπαίθρου εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Μέχρι στιγμής είχαμε ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης υπαίθρου με το οποίο, ε, αν θέλετε, συμβίωναν και όλες αυτές, και όλα αυτά τα 16 σχέδια. Τώρα όμως δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ε, του εθνικού σχεδίου που θα συνυπάρχει με τα περιφερειακά. και όταν υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία ε, θα μπορούσαν να ευνοήσουν πολλές περιφέρειες ταυτόχρονα, δυστυχώς δεν μπορούμε να εκπονήσουμε ένα σχέδιο ενιαίο πλέον. Καλό θα ήταν λοιπόν να μπορεί στο άρθρο 7 να συμπεριληφθεί μια πρόταση που θα λέει ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα σχέδιο για τη χρηματοδότηση διαπεριφερειακών σχεδίων ή προγραμμάτων. Τέλος, ένα θέμα που θέλω να υπογραμμίσω και το οποίο θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι οι αγρότες θα μπουν σε κάποιες οργανώσεις παραγωγών. Όταν έχουμε οργανώσεις παραγωγών όμως που έχουν κάποια δύναμη και ε, ισχύ, αυτές θέλουν να τις περιορίσει η Κομισιόν. Άρα δεν είναι η πρόταση αυτή σωστή. Επίσης θα πρέπει η... Ε, βοήθειες που δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να ε, περιοριστούν τελικά. Γιατί λέμε ε, θέλουμε να έχουμε συγχώνευση, ομαδοποίηση παραγωγών. Βλέπω ότι ο Γάλλος συνάδελφος νεύει καταφατικά. Μετά λέμε ότι πρέπει να βοηθούμε τις ΜΜΕ. Πώς θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Και τέλος να πω ότι σε αυτή την πρόταση του κυρίου Κάπουλας για την ανακατανομή των κεφαλαίων του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα δεν μπορώ να συμφωνήσω. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω γιατί η πολιτική συμφωνία αφορά μόνο ε, τον πρώτο πυλών. Όχι, δεν μιλώ μόνο για τη συμφωνία του Συμβουλίου, αλλά μιλάω και για την έκθεση του κυρίου Άλμπερτ Ντες. Το καλοκαίρι συγκεκριμένα, όταν ψηφίσαμε, είπαμε ότι θα πρέπει να αναφέρει, να αφορά τον πρώτο πυλώνα αυτή η αναδιανομή και νομίζω ότι αφού έχουμε λάβει αυτή την απόφαση πρέπει να την τηρήσουμε, να τη σεβαστούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ράνθ. Κώστην και να πω Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ισηγητά για τις παρουσιάσεις σας και για κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις που κάνατε. Θα ήθελα να ε, τονίσω πόσο σημαντικό είναι ε, να εξετάσουμε όχι ξεχωριστά τον πρώτο από τον δεύτερο πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά να έχουμε η υπόψη μας πάντα την ε, σχέση μεταξύ τους. Ιδιαίτερα το πρόγραμμα γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων στον δεύτερο πυλώνα είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά το screening στον πρώτο πυλώνα, έχουμε χώρες στην Ευρώπη που έχουν κάνει πολλά στον ε, τομέα των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων τις τελευταίες δεκαετίες και θα πρέπει να αποκλείσουμε το greening που προτείνεται, το πρασίνισμα, να αποτελέσει οπισθοδρόμηση της περιβαλλοντικής γεωργίας σε πολλά κράτη-μέλη. Και θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν στην οικολογική γεωργία να μπορούν να συμπεριληφθούν και στο greening, το πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας εδώ και ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Τα μέτρα για το πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα είναι μονοετή. Όταν εκμεταλλεύσεις συμμετέχουν στο πρασίνισμα, μιλάμε για πολυετή μέτρα. Η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα λοιπόν είναι πολύ σημαντικές εδώ. Τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα έχουν αποδείξει την αξία τους και στις περιπτώσεις όπου έχουμε ε, αφήσει στα κράτη-μέλη τις αποφάσεις ε, βλέπουμε σημαντική πρόοδο. Θα πρέπει να ληφθούν οι υπόψη οι διαφορές ανάμεσα στα διάφορα Θα ήθελα να ε, τονίσω ότι όσον αφορά τις εταιρικέ σχέσεις, ε, τη, ε, τη σχέση ανάμεσα στα διάφορα ταμεία, θα είναι σημαντικό να αποφύγουμε τις διπλές χρηματοδοτήσεις, ωστόσο θα πρέπει στα πλαίσια των συμφωνιών εταιρική σχέσης να αποφύγουμε την αύξηση της γραφειοκρατίας για τα ταμεία αυτά. και να αποφύγουμε και τα πολιτικά παιχνίδια στα κράτη-μέλη ε, όσον αφορά την ε, χρήση των πόρων αυτών. Ο εισηγητής ήδη το είπε. Ε, θα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και θα είναι απαραίτητες και είναι απαραίτητα τα στοιχεία της Κομισιόν, τα οποία όμως είναι ελλειπή. Ε, ο κ. Ε, στην έκθεσή του έχει αναφέρει το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε στα τυφλά να λαμβάνουμε αποφάσεις όταν δεν ε, είμαστε πεπισμένοι ότι θα είναι προς όφελος των μειονεκτικών περιοχών. Θα πρέπει να εξετάσουμε τα αντισταθμιστικά μέτρα για τις ορεινές περιοχές. Επικροτούμε τις προτάσεις που γίνονται για τον τομέα αυτό. Σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την ύπεθρο. Ε, τα μέτρα αυτά όμως δεν θα λειτουργήσουμε αν δεν προσέξουμε και την κτηνοτροφία. Θα πρέπει και αυτή να συμπεριληφθεί στον κανονισμό. Κεντρικά ε, σημεία το, της πρότασης είναι η επενδύσεις, η εκπαίδευση, η κατάρτιση. Χρειαζόμαστε από πλευρά της Κομισιόν ε, συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή. Οι εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικές. Χρειάζονται λοιπόν κατάλληλες ε, συνθήκες ε, πλαισίου. Ο συνάδελφος ήδη αναφέρθηκε στους νέους γεωργούς. Τα μέτρα που προτείνονται στον πρώτο πυλώνα δεν αρκούν καθόλου για ένα πρόγραμμα και για τους νέους γεωργούς. Χρειάζονται πολύ συγκεκριμένες περαιτέρω προτάσεις, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά την υποστήριξη κατά ε, την ε, την έναρξη επαγγέλματος των νέων γεωργών, την, την απόκτηση μιας εκμετάλλευσης. Επίσης, όσον αφορά την βιομάζα, υπάρχει εδώ σημαντικό δυναμικό για τις εκμεταλλεύσεις μας και είναι και εδώ ο παράγοντας θέσης απασχόλησης ε, σημαντικός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μάρτιν Όσλιν. Ε, ναι, ο κύριος Κάπουλας έχει απόλυτη το δίκιο. Ε, στην πρόταση της Κομισιόν υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες ε, στις οποίες θα θέλαμε να απαντήσει. Οι στόχοι είναι σωστοί, αυτοί που αναφέρονται, αλλά ε, σημαντικό ερώτημα είναι όταν θέλουμε περισσότερη ευελιξία σχέση με άλλα προγράμματα και τα ταμεία, μήπως θα είναι αυτό η βάρος της υπαίθρου, μήπως η παραμερίζεται για να δοθούν αλλού τα χρήματα. Δεν είναι απλό το θέμα αυτό. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην, παραμείνει ανεξάρτητη η ανάπτυξη της υπαίθρου. Σημαντικό ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί είναι η συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων στον δεύτερο πυλώνα. για πολλά κράτη-μέλη θα είναι σημαντικό πρόβλημα η συγχρηματοδότηση των ε, προγραμμάτων αυτών. Ή θα πρέπει να αλλάξουμε το πλαίσιο ώστε να θέσουμε προτεραιότητες όπου θα δώσει περισσότερους πόρους η Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα καταλήξουμε στην ε, περίπτωση να έχουμε πολλά καλά προγράμματα, τα οποία όμως να μπορούν να εφαρμοστούν, διότι δεν θα μπορούν τα κράτη-μέλη να συγχρηματοδοτήσουν. Εδώ θα πρέπει να δοθεί απάντηση. Όσον αφορά το σχέδιο της Κομισιόν, αναφέρεται το ποσοστό του 25% για τα περιβαλλοντικά μέτρα του δεύτερου πυλώνα. Εδώ όμως υπάρχει κάποιο έλλειμμα. Θα πρέπει να φροντίσουμε τουλάχιστον το 25% για τα περιβαλλοντικά μέτρα στο δεύτερο πυλώνα να διατηρηθεί αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Έχουμε θέσει τους ε, στόχους στον ε, πρώτο πυλώνα, αλλά η περιβαλλοντοποίηση το ε, αναφέρεται και στον δεύτερο πυλώνα. Και τέλος, θα πρέπει να προσέξουμε τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα στην Ευρώπη. να είναι δεσμευτικά σε κάποιο βαθμό σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ε, διαφορές όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο ε, ανάλογα με τις χώρες. Ο συνάδελφος από την ε, Αυστρία ανέφερε σωστά ότι η Αυστρία έχει αναπτύξει πολύ τους τομείς του δεύτερου πυλώνα θετικά για την Ήπεθρο, ενώ υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη όπου δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Θα πρέπει να πετύχουμε ισορροπία εντός Ευρώπης. Όσον αφορά τις μειονεκτικές περιοχές, ε, σημαντικό είναι να ε, μπορούν να λάβουν τους πόρους. Ε, βρίσκω λάθος όμως να συζητήσουμε ταυτόχρονα το θέμα της νέας οριοθέτησης καθώς και της χρηματοδότησης. Θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός των δύο αυτών θεμάτων. Εάν συζητάμε την νέα οριοθέτηση ταυτόχρονα με την οικονομική ενίσχυση, αυτό θα είναι λάθος. Ε, έχω πει ότι κατά τη γνώμη μου κάποια θέματα δεν εμπίπτουν στον δεύτερο πυλώνα. Η ιδιωτική ασφάλιση στον γεωργικό τομέα δεν πιστεύω ότι πρέπει να ε, συγχρηματοδοτείται. Δεν αποτελεί αυτό ε, θέμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε στενά πλαίσια. Ε, δεν θα πρέπει εδώ να ε, ασχολούμαστε με διαχείριση του κινδύνου στον τομέα των ιδιωτικών ασφαλιών και να δημιουργούμε σχετικά ταμεία. Αυτό αποτελεί λάθος προσέγγιση. Γενικά, θα πρέπει και πάλι να πω στον, ε, στον εισηγητή ότι έχει δίκιο ε, θα πρέπει να δούμε πού θέλουμε να δώσουμε χρήματα και ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον δεύτερο πυλώνα στις συζητήσεις ε, στο ίδιο επίπεδο με τον πρώτο βαθμό. οικονομικά όμως δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να γίνουν περικοπές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μάρτιν ή κυρία Ρόντουστ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι με τις προτάσεις ε, του Λουίς ε, Καπουλασάντος. Ε, νομίζω ότι πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση για μένα είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι χρειαζόμαστε, ε, συνεχίζουμε να χρειαζόμαστε έναν, δεύτερο, έναν ισχυρό δεύτερο πυλώνα. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μένουν στην Ήπεθρο και θα, είναι, θα πρέπει να τους δείξουμε πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη ε, πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη και για τους ανθρώπους και πόσο μάλλον στην ε, Ήπεθρο. Χρειαζόμαστε τους αντίστοιχους πόρους και αν η Κομισιόν ε, δεν ε, έχει καθορίσει τα ποσά, ίσως ε, θα πρέπει εμείς να αναφέρουμε συγκεκριμένα ποσά και θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε κάτι με τα χρήματα αυτά. Στο μέλλον τα τρία βασικά ευρωπαϊκά ταμεία θα εξετάζονται από κοινού, αυτό το βρίσκω χρήσιμο. Σημαντικό όμως για μένα είναι το παλιό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπέθρου να το διαχειριζόμαστε εμείς και εμείς να μπορούμε να ε, ορίσουμε για ποια μέτρα, για ποια προγράμματα θα ε, δίδονται τα χρήματα. Σημαντικό είναι επίσης να σκεφτούμε να μην έχουμε αποκλειστικά πόρους για συγχρηματοδότηση στον κανονισμό αυτό, διότι ξέρω ότι υπάρχουν και οι ιδιώτες που έχουν ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με την πρόθεση της ε, ανάπτυξης της υπαίθρου. Επίσης, ε, σημαντικό είναι να σκεφτούμε μήπως ε, η ε, εργασία χωρίς αμοιβή μπορεί να θεωρηθεί ε, συγχρηματοδότηση. Να εξετάσουμε δηλαδή και άλλους τρόπους συγχρηματοδότησης χωρίς μετρήτα. Μήπως θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε και τη συμπερίληψη του ΦΠΑ εδώ σημαντικά προβλήματα ε, έχουμε όσον αφορά την, ε, τον καθορισμό των ε, μειονεκτικών περιοχών. Κατά τη γνώμη μου, ο ορισμός και τα κριτήρια τα οποία έχει υπαγορεύσει το ελεκτικό συνέδριο δεν είναι σκόπιμοι. Υπάρχουν περιοχές που έτσι μπορούν να θεωρηθούν προωθούν μειονεκτικές που κατά τη γνώμη μου είναι από τις ε, πιο πλούσιες σε κάποιους πόρους. Ε, για παράδειγμα οι υδροβιότοποι, η βάλτη Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου. Ευχαριστώ πολύ. Μισελ Νταντά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για την ε, παρουσίασή του. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει κάποιες επιλογές στο δεύτερο πυλώνα. Προτείνει κονδύλια για την καινοτομία, για την ε, ατομική διαχείριση των συμβάσεων δίνει μια πιο σαφή θέση στα δάση και τις μη ευνοημένες περιοχές, ε, ορεινές περιοχές κτλ. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν ε, οι επιθυμίες όλων. Άρα πρέπει να γίνουν κάποιες επιλογές. Η Επιτροπή μας έχει συζητήσει μεταξύ άλλων ε, το θέμα της ανανέωσης των γενεών αν λάβουμε υπόψη μας και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η πέθρος αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία, αλλά δεν τα εφαρμόζουν ε, οι χώρες. Εξού και έχουμε 6% ε, μείωση της ε, εκμετάλλευσης. Είναι ένα θέμα λοιπόν που είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την παραγωγή και σήμερα, αλλά και για το μέλλον. Μήπως λοιπόν τα μέτρα υπέρ τη εγκατάστασης θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικά, Υποχρεωτικέ εφαρμογέ για όλες τις χώρες. Ξέρω ότι είναι πολύ ευκολότερο ένας ε, αγρότης ε, να ε, δει τον γείτονά του να κλείνει το, την εκμετάλλευσή του και έτσι αυτός να παίρνει τη θέση του παρά να βλέπει ένα νεαρό αγρότη να έρχεται δίπλα του ως ανταγωνιστής. Αλλά εκεί θα έπρεπε να δώσουμε την προσοχή μας ό,τι αφορά την ορεινή γεωργία κάνει μια καλή πρόταση η Κομισιόν, δηλαδή μεγαλύτερους πόρους να δοθούν, σε περίπτωση υπάρχει κάποιο φυσικό ε, μειονέκτημα, ως αντιστάθμιση δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε στην Κομισιόν ότι εδώ και πολλούς μήνες ζητούμε από την Κομισιόν να μας δείξει τους χάρτες που μεταφράζουν στην πράξη την πρόταση κανονισμού της. Είναι ένα αίτημα το οποίο είχε διατυπώσει ο συνάδελφος Ντόρφμαν στην έκθεσή του πριν από αρκετούς μήνες δεν ξέρω αν δεν έχω καλή ενημέρωση, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω δει ποτέ τους χάρτες αυτούς. Αλλά μιλάμε για μια συζήτηση πάρα πολύ σημαντική. Και σίγουρα βαραίνει η συζήτηση του τι θα γίνει με την ΚΑΠ στην όλη αυτή εκστρατεία, αλλά και σε αυτό θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Η σχέση τώρα με τις κοινέ οργανώσεις αγοράς. Υπάρχουν ε, κάποια κεφάλαια με τα οποία θα μπορούσαν να ε, δημιουργηθούν ισχυρές ενώσεις παραγωγών και κοινέ οργανώσεις αγοράς. Και προτείνει στις οργανώσεις παραγωγών να βάζουν κάποια ε, κονδύλια κατά μέρος και όταν δεν είναι καλή εσοδεία να μπορούν να διατεθούν και βάζει και κάποια, κάποια ποσά εκεί. Επειδή είναι ένα θέμα πολύ λεπτό, νομίζω ότι θα πρέπει να το επεξεργαστούμε από κοινού. Γιατί πολλές φορές οι αγορές ε, κυμαίνονται, έχουν διακυμάνσεις. Το να έχουμε ένα συλλογικό εργαλείο στα χέρια των οργανώσεων παραγωγών νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. στην κοινή οργάνωση αγοράς ούτε για τα φρούτα ούτε για, γάλα, για το γάλα είδαμε να το αξιοποιούν. Ευχαριστώ. Έμερες και μετά Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή που ζήτησε τη συμβολή μας για την έκθεση που θα γράψει. Σήμερα ακούσαμε ήδη πολλές προτάσεις. Θα ήθελα όμως να αναφέρω ότι πρέπει να πετύχουμε και τη σωστή στάθμιση ανάμεσα στους διάφορους τομείς του δεύτερου πυλώνα. Διότι πέρα από περιβαλλοντικά προγράμματα θα χρειαστούν και επενδυτικά προγράμματα και θα πρέπει να εξετάσουμε και τη διαφορετική ανάπτυξη της υπαίθρου, ε, ιδιαίτερα αν εξετάσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Χρειαζόμαστε ανθρώπου ε, στην Ήπεθρο, αλλιώ ε, θα νιώθουν πολύ μοναχικά εκεί. Στο μεταξύ όμως ε, θα πρέπει και τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο. Έχουμε λοιπόν εδώ σημαντικά καθήκοντα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει η σωστή γιατρική περίθαλψη. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, δεν θα πρέπει να τα ξεχάσουμε διότι θέλουμε να ε, προωθήσουμε την ανάπτυξη της υπαίθρου. Επίσης ε, με το κοινωνικό, το ε, ταμείο, το αλληλευτικό ταμείο και το διοργικό θα πρέπει να πετύχουμε καλές διασυνδέσεις και θα πρέπει να εξετάσουμε πιθανούς τρόπους συγχρηματοδότησης. Για παράδειγμα, για τα, προγράμματα, για τα επενδυτικά προγράμματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία, τα οποία να διαχειρίζονται μεγάλες περιφερειακές ε, τράπεζες ε, ώστε να ε, μπορούμε να έχουμε περισσότερες δυνατότητες σε πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων. Μπορούμε να πετύχουμε εξωτερική ανάθεση εφόσον χρησιμοποιούμε ήδη γνωστές τράπεζες και θα πρέπει να επιτρέπουμε να υπάρχει και κάποιος κίνδυνο ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε νέες ιδέες και θα πρέπει να σκεφτούμε μήπω θέλουμε και ε, έναν ε, μηχανισμό ε, εξοικονόμηση εξοικονόμησης αποταμίευσης ώστε να μπορούμε να πετύχουμε την πολλαπλή χρήση διάφορων πόρων ώστε να μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Ε, Όπω και όλοι οι άλλοι, πάντω προσβλέπω στη συνέχιση των καλών συζητήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπρίτα. Κυρία Καρνιέτε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πάμε πίσω λίγα χρόνια, το 2008, όταν η Λετωνία αντιμετώπισε μια πολύ βαθιά οικονομική κρίση. Η Λετωνία είναι μια χώρα 2 εκατομμυρίων και λόγω αυτής της κρίσης γύρω στις 200.000 άνθρωποι έφυγαν από την Λετωνία για να αναζητήσουν δουλειά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή το 1 δέκατο του πληθυσμού μας. Αυτοί που έφυγαν είναι από τις νεότερες, νεότερη γενιά και κυρίως από γεωργικές περιοχές. Γι' αυτό για τη Λετωνία δεν είναι μόνο θέμα ανάπτυξης, αλλά και θέμα εθνικής ασφάλειας η ανάπτυξη της υπαίθρου. Διότι οι συνοριακές μας περιοχές, οι παραμεθόριες περιοχές είναι σχεδόν κενές και οι παραμεθόριες μας περιοχές είναι και οι συνοριακές περιοχές της επικράτειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρήματα στα οποία βασίζεται η Λετωνία είναι αυτά που προέρχονται από τα διευθυντικά ταμεία και από την ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι τα μόνα χρήματα που μπορούμε να βάλουμε στην ανάπτυξη και που μπορούν να φέρουν ανάπτυξη και να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης στις περιοχές της υπαίθρου. Εγώ Εκτιμώ ε, πολύ την ιδέα του εισηγητή να αναζητήσουμε χρηματοδότηση στην πρώτη και δεύτερο πυλώνα από κοινού. Ε, στην περίπτωση της ε, Λετωνίας δεν αλλάζει και πολύ, γιατί αν συνδυάσουμε τα κονδύλια αυτά ε, και πάλι παίρνουμε λιγότερα από όλες τις υπόλοιπες 26 χώρες. Αυτό που με ανησυχεί ωστόσο είναι ότι αυτοί οι δύο πυλώνες έχουν διαφορετικούς στόχους. Η ανάπτυξη η αγροτική και για τη χώρα μου και πιστεύω για όλες τις χώρες είναι πολύ μεγάλη σημασία και μας ενδιαφέρει στην επόμενη περίοδο γιατί τα κριτήρια του δεύτερου πυλώνα ε, έχουν εδώ αναθεωρηθεί. Εμάς μας ανησυχεί η ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά εγώ θα ήθελα να μιλήσω και για την αλλαγή των γενεών. πριν από λίγα χρόνια ήμασταν τυχεροί γιατί το 18% των γεωργών μας ήταν νεότεροι κάτω των 35 ετών. Λόγω αυτής της μαζικής μετανάστευσης, οι τελευταίες μας στατιστικές δείχνουν ότι γύρω στα 6% είναι πια κάτω των 35 ετών. Γι' αυτό και η Λετωνία στηρίζει εντόνως τις ιδέες για ενίσχυση της προσβασιμότητας στη γη για νέους αγρότες, για εξοπλισμό, για κεφαλοποίηση και για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είμαστε 27 διαφορετικές χώρες με 27 διαφορετικές ε, γεωργικές δομές και γι' αυτό το στοιχείο της ευελιξίας στο δεύτερο πυλώνα είναι σημαντικό. Αλλά πιστεύω ότι για κάθε μέλος της Επιτροπής Γεωργίας η μεγαλύτερη ανησυχία είναι Τελική απόφαση για το συνολικό προπολογισμό. Ποιο θα είναι το τμήμα των κονδυλίων που θα δοθεί στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα. για την γεωργία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αντέξουμε την περικοπή των πόρων και ότι θα έχουμε ανθίζουσες ορτικές περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καλνιέτε. Ο Αντιπρόεδρος Σικέρσκι και μετά η κυρία Κάντενμπακ. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να διερωτηθούμε την ίδια ερώτηση, δηλαδή τι είναι η γεωργική ανάπτυξη γενικά. Πρόκειται για επιχειρηματικότητα, νέες θέσεις, υποδομές, περιβαλλοντική προστασία, βιοπικιλότητα ή πρόκειται για την ανάπτυξη αγροκτημάτων ή πρόκειται για καινοτομία ίσως. Ίσως για ψηλότερα εισοδήματα. Η δεύτερη πυλώνας αφορά τις επενδύσεις. Η άρδευση μπορεί εδώ να ε, παίξει αποφασιστικό ρόλο στο μέλλον όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Εγώ βλέπω κάποια προβλήματα. Θα ήταν καλή ιδέα να χρησιμοποιήσουμε την ιδέα της Επιτροπής για να λάβουμε υπόψη κάποια ποιοτικά κριτήρια, αέπανα κατά κεφαλήν, διότι πρόκειται για υποστήριξη κάποιων λιγότερο ευνοημένων περιοχών. Δεν ξέρω πώς να ερμηνεύσω την πρόταση του εισηγητή για συγχώνευση των δύο πυλώνων, γιατί οι δύο πυλώνες παίζουν διαφορετικό ρόλο και έχουν διαφορετικό στόχο. Ο πρώτος αφορά όλους τους γεωργούς, ενώ ο δεύτερος μόνο αυτούς που συμμετέχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα για τις περιοχές της Πέθρου. Θα ήταν δύσκολο να ε, συνδυάσουμε τους δύο πυλώνες. Κάτι ακόμα, μιλάμε για βιοπικιλότητα πολύ συχνά και η εντύπωση μου είναι ότι η βιοπικιλότητα χρησιμοποιείται από αυτού που θέλουν ε, γρήγορα να μεταρρυθμιστεί η ΚΑΠ. Θα πρέπει να εστιάσουμε στη βιοπικιλότητα και να χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση ενός κοινού γεωργού και όχι ε, από την προσέγγιση αυτών που θέλουν γρήγορα τα χρήματά τους. Ένα άλλο θέμα είναι η πολιτική για την ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα. Σε ποιο βαθμό θα πρέπει αυτό να συνδέεται με την πολιτική συνοχής. Διότι η πολιτική πολιτική συνοχή ε, μπορεί να στηρίξει μεγάλα αστικά κέντρα που είναι τα κέντρα καινοτομία και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Όταν όμω μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, δεν μπορούμε να ξεχνάμε την ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Ας μην ε, χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες αρχές όπως αυτές για την γεωρική πολιτική σε όλα τα κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο. Η συνάδελφος μίλησε για τις περιφέρειες. Πράγματι, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Μιλήσατε επίση ε, για κάποια ποσοστά, 50 για το ένα, 20 για το άλλο, 25% για το τρίτο. Όχι, δεν μιλάμε ε, για αυτό και θα ολοκληρώσω. Ε, η κυρία Καλνιέτε δεν μίλησε γι' αυτό. Η κυρία Καλνιέτε είπε κάτι πολύ σημαντικό. Εντάξει, μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώ ποια θα είναι τα κονδύλια, ποιο θα είναι ο προπολογισμό, γιατί είναι υπό επεξεργασία αυτή τη στιγμή, αλλά Μπορεί να γίνουν κάποιε αλλαγέ, ότι κόβεται ένα κονδύλι από εδώ, πάει κάπου αλλού. Τι θα γίνει στην προκειμένη περίπτωση, από πού θα κοπούν οι πόροι από την κοινή γεωργική πολιτική, από τον πρώτο πυλώνα, από τον δεύτερο πυλώνα. Σα τα λέω αυτά γιατί μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Και καλό θα είναι να έχουμε σκεφτεί κάποιε πιθανέ λύσει, να τι συζητήσουμε εδώ, να δούμε όλα αυτά τα σημεία τα οποία είναι σημαντικά και θα πρέπει και με τις κυβερνήσει μα σε εθνικό επίπεδο να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Σικέρσκη και τώρα το λόγο έχει η κυρία Κάντερμπακ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή Καπλά ε, Είμαι ε, εισηγήτρια ε, στην άκρη και στην ΕΝΒΗ. Είναι πολύ καλό να έχουμε εδώ έναν καλό εισηγητή διότι υπάρχουν Φυσικά διαφορετικές απόψεις ε, στις διάφορες επιτροπές ε, και οι συζητήσεις έχουν δείξει ότι ο πρώτος ε, πυλώνας είναι ο πιο επίκαιρος, ενώ ο δεύτερος πυλώνας, η ανάπτυξη της υπαίθρου, προσανατολίζεται περισσότερο στο μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εδώ να παίξει ένα σημαντικό ρόλο από πλευράς του Συμβουλίου. Ε, υπάρχει, ασκείται σημαντική πίεση όσον αφορά τον ε, πρώτο πυλώνα, τις άμεσες πληρωμές, ε, ενώ τα καθήκοντα που σχετίζονται με τον δεύτερο πυλώνα είναι πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τα όρια της συγκεκριμένη θητείας. Δεν είναι λοιπόν πάντα εύκολο ε, στα διάφορα κράτη-μέλη να ε, διατεθούν οι πόροι. Έτσι λοιπόν ε, συχνά τα περισσότερα χρήματα, κινδυνεύουμε τα περισσότερα χρήματα να δοθούν στον πρώτο πυλώνα και ο δεύτερος πυλώνας να θεωρηθεί περισσότερο μια προσθήκη, ένα συμπλήρωμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Κάτεμπακ. Τώρα με Μίτσακ και μετά Νεντελτσέβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί νομίζω ότι έχει πραγματικά μπει σε πολλή λεπτομέρεια ε, αναλύοντας την πρόταση της Κομισιόν. Έχω διάφορα σχόλια. Πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε ο δεύτερος πλέον είναι στο δυνατόν ε, πιο κοινοτικό. Ε, όταν μιλάμε δηλαδή για επενδύσεις ε, στον τομέα τη μεταποίησης κτλ. Θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε υπό την προοπτική της όλης Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινότητας εν γέννη. Σήμερα είναι έτσι η κατάσταση που κάποιοι αγρότες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια για την έρευνα, ενώ κάποιοι άλλοι μπορούν. Η κατάσταση δεν είναι δίκαιη για παράδειγμα, για την δημιουργία ενός θερμοκηπίου μπορεί κάποιος να πάρει χρήματα σε μια περιοχή ενώ σε κάποια άλλη περιοχή να μην μπορεί να πάρει. Αυτό λοιπόν καταστρέφει τον ανταγωνισμό. Το ίδιο ισχύει και με τον τομέα της μεταποίησης. Επομένως νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ε, εστίαση στο κοινοτικό σκέλος και μεγαλύτερη χρήση της κοινοτική μεθόδου. Δεύτερο θέμα. Ο δεύτερος πυλώνας νομίζω ότι θα πρέπει να ε, αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη αλλά πάρα πολύ προσεκτικά θα πρέπει να κινηθούμε. Το έχουν και οι προλαλήσαντε. διότι σε ορισμένες περιφέρειες Έχουμε υπερβολικέ επενδύσει. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά κονδύλια που διατίθενται στι επενδύσει. Άρα, το αποτέλεσμα είναι πλεόνασμα στην παραγωγή. Και έτσι θα πρέπει να υπάρξει ένα έλεγχο ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτά τα επίπεδα. Κάτι άλλο που νομίζω ότι λείπει από τις αποφάσεις μας είναι το εξή. Νομίζω ότι είναι κοινό γνωστό ότι και στην Πολωνία αλλά και σε άλλε χώρε πολλοί πόροι, πάρα πολλοί πόροι έχουν ταπανηθεί για μέτρα τα οποία τελικά αποδείχθηκαν υπερβολικά ή είχαν ως αποτέλεσμα να αγοραστούν υπερβολικά πολλά μηχανήματα για τον τομέα της μεταποίησης ή να μην είναι σωστά τα σωστά μηχανήματα αυτά που αγοράστηκαν και ούτω καθεξής. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα για το μέλλον. Η βιοπικιλότητα είναι ένα άλλο θέμα επίσης, η προστασία της φύσης. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει λύσεις να αναζητηθούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την ευελιξία, πρέπει νομίζω να διατηρηθεί η ευελιξία για τα διάφορα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές, διαρθρωτικές αποφάσεις. Διότι η κατάσταση από τη μια χώρα στην άλλη διαφέρει. Και θα πρέπει να σταματήσει η αστιφιλία να ε, αρχίσει ο κόσμος να επιστρέφει στην Ήπεθρο γιατί την θεωρεί ε, ελκυστική. Θα πρέπει επίσης να περιορίσουμε κάποιες τον, αριθμό των εκμεταλλεύσεων των γεωργικών και να δημιουργήσουμε τις ε, σωστές συνθήκες με την παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης για αυτούς που θέλουν να αλλάξουν τρόπο ζωής. Θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα επίπεδα παραγωγής στους διάφορους τομείς. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν κάποια ευελιξία. Θα πρέπει να βλέπουμε την κατάσταση χωριστά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Τέλος, επενδύσεις στην Ήπεθρο. Νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά με αυτούς που ασχολούνται με την πολιτική συνοχής ώστε να δαπανούνται στον δυνατόν πιο αποτελεσματικά τα κονδύλια. Όταν μιλάμε για τις δημόσιες υπηρεσίες, τις υποδομές, την, ε, το χτίσιμο σχολείων, την υγειονομική περίθαλψη κτλ. Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες διαφορές στο επίπεδο και την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών μεταξύ υπαίθρου και αστικών κέντρων. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε κάποιους πόρους και από τα ταμεία συνοχής. Μάλιστα. Τώρα η Μαρία Νεντελτσέβα και μετά Φέλτερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κάπουλα Σάντος και να πω ότι ναι πράγματι πρέπει να καθορίσουμε τους κοινού μα στόχους. Επίσης σημαντικό είναι να διδαχθούμε από την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα. Αν με επιτρέπετε θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα που αφορούν συγκεκριμένα τη Βουλγαρία. Πρώτα απ' όλα, τα μέτρα για τον δασικό τομέα. Το χρηματοδοτικό μέσο για τον τομέα αυτό είναι το Εθνικό Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη των Ζωνών της Υπαίθρου και περιλαμβάνει μέτρα τα οποία μας επιτρέπουν να προστατεύσουμε τα δάση μας και να εξασφαλίσουμε μια αηφόρο διαχείριση. Ωστόσο, η Βουλγαρία είναι μια χώρα όπου το 76%, πάνω μάλιστα από το 76% των εκτάσεων, των εκτάσεων είναι κρατικές. Αυτό το ποσοστό που είναι τόσο ψηλό δεν μας επιτρέπει να ζητήσουμε στήριξη, ενίσχυση στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ε, ενίσχυσης ε, των ε, αγροτικών ζωνών. Δεν είναι λοιπόν αποτελεσματικό αυτό το πρόγραμμα για εμάς και επομένως δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα που χρειάζονται ούτε και να απορροφήσουμε τους πόρους που μας είναι αναγκαίοι. Δεδομένης της μεγάλης σημασίας του δασικού τομέα για την Ευρώπη συνολικά, νομίζω ότι είναι αναγκαίο τα μέτρα τα οποία προβλέπονται για τα δάση να έχουν ένα μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής ώστε να μπορούν να περιλαμβάνονται και οι κρατικές δασικές εκτάσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαχείριση των κινδύνων, θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπαν οι συνάδελφοι. Υπάρχουν διάφορα μέσα στα οποία για τα οποία, τα οποία μάλλον διέπονται από τα άρθρα 68, 70 και 71 του κανονισμού. Θα πρέπει, πιστεύω, να λάβουμε υπόψη μας και νέα μέτρα και ε, καινούργιες διατάξεις διαχείριση των κινδύνων. Να πούμε επίση ότι η βοήθεια παρέχεται σε λίγα κράτη-μέλη και πολλές φορές υπάρχει σε ένα τέλος διαφορετικό εκτός του τομέα της γεωργίας σύστημα τους αγρότες. Έχουμε τους όρους του άρθρο 68. Δεν νομίζω ότι αντικατοπτρίζονται στο νέο πακέτο των μέσων διαχείρισης ε, κινδύνου. Επομένως, το μόνο που θα κάνουμε νομίζω είναι να περιπλέξουμε τις διαδικασίες και όχι να τις απλουστεύσουμε. Ούτε θα απαλύνουμε το διοικητικό άχθος. Άρα θα δημιουργήσουμε ένα ακόμη πρόβλημα για τους αγρότες. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει ένας πιο αποτελεσματικός έλεγχος στα κρατημέλη. Θα ήθελα να αναφερθώ και λίγο και στις επενδύσεις στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή. Να περιληφθεί δηλαδή και η κτηνοτροφία. Γιατί για την Βουλγαρία αυτό είναι ένα θέμα πολύ συγκεκριμένο. Νομίζω ότι η κτηνοτροφία, ένα τομέα κλειδί, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να είναι και στο επίκεντρο της δικής μας προσοχής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το 5% που προτείνει η Κομισιόν, για να εγγυηθεί την πιο αποτελεσματική εφαρμογή. Αυτό το ποσοστό του 5% ε, μας βρίσκει σύμφωνος. Αυτό το 5%, αυτός ο μηχανισμός όμως με το 5% μήπως τελικά επιβαρύνει και μήπως προκαλέσει νέες διαδικασίες διοικητικές. Μήπως τελικά τα κριτήρια του ελέγχου δεν, ε, γίνουν, δεν καταστήσουν ακόμη πιο δύσκολους τους ελέγχους. Αντί δηλαδή να διευκολύνουμε τα πράγματα, μήπως δημιουργήσουμε νέα εμπόδια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 έχει θέσει ως στόχο της το 20% όλων ε, των ευρωπαϊκών πόρων ε, να διατεθεί για την ε, καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το κείμενο που έχουμε μπροστά μας όμως δυστυχώς δεν φροντίζει το 20% του Ταμείου για την Ανάπτυξη της Υπέθρου να χρησιμοποιηθεί για τους όρους αυτούς. θα πρέπει να ε, επικεντρωθούμε στην ε, απόδοση της ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να πετύχουμε το στόχο μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, διότι η γεωργία κατά την παραγωγή τροφίμων παίζει σημαντικό ρόλο εδώ. Ε, η γεωργία καταναλώνει πολύ ενέργεια. Ο συνάδελφος Σεμποβή ήταν αρμόδιος για το θέμα αυτό και έχει περιγράψει αναλυτικά την αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας. Είναι σημαντικό να βρούμε πιο αποτελεσματικές λύσεις για την κατανάλωση της ενέργειας και για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν σε μεγάλο ποσοστό ε, να χρησιμοποιηθούν ε, στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να στηρίξουμε όχι όμως μόνο ε, την γεωργία και την παραγωγή ενέργειας, θα πρέπει να στηρίξουμε και τους δήμους, τα σχολεία και είναι αυτοί οι οργανισμοί που μπορούν να λαμβάνουν, να τροφοδοτούνται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για παράδειγμα, για τη θέρμανσή τους. Πιστεύουμε ότι και εδώ θα πρέπει να ε, παράσχουμε την υποστήριξή μας. Ε, επίσης, ε, χρειαζόμαστε εγκαταστάσεις άρδευσης ε, στην Ευρώπη. Θέλουμε να διαμορφώσουμε καλύτερα την Ήπεθρο. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Ζητώ συγγνώμη από τον εισηγητή που δεν ήμουν στην αίθουσα από την αρχή. Θέλω να θίξω δύο θέματα. Το ένα αφορά τα άρθρα 29 και 30 για την γεωργία που είναι φιλική προς το περιβάλλον. Θα πρέπει να ζητήσουμε από σαφήνιση από την Κομισιόν για το πώς αυτό σχετίζεται με το πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα. Δεύτερη μου παρατηρήση αφορά μια ενδιαφέρουσα ιδέα που και πάλι όμως δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες που είναι οι ευρωπαϊκές εταιρικέ σχέσεις για την καινοτομία. Οπότε ό,τι κατάλαβα στη τελευταία μεταρρυθμίση και αυτό ήταν θέμα. Δεν κατάλαβα όμως τι έγινε στα κράτη-μέλη, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ποιε είναι οι διαφορέ, Αλλά σίγουρα εγώ υποστηρίζω την ιδέα του να έχουμε ένα πολύ καλό συμβουλευτικό σύστημα. Νομίζω πω η ανησυχία των ε, Γεωργών ήταν ότι ένα προπολογισμό που παραδοσιακά θα πήγαινε σε εκείνου για ε, διαρθρωτικά μέτρα και ανταγωνιστικά μέτρα θα ε, απορροφηθούν από το συμβουλευτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να πάρουμε περισσότερε λεπτομέρειε από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Grazie adesso la parola Ευχαριστώ. Τώρα έχει το λόγο ο Αντιπρόεδρος Βοτσιχόφσκι. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Πρασίνισμα της ε, γεωργικής οικονομίας, πρώτος και δεύτερος πυλώνας. Η πρόταση της Κομισιόν αφορά νέες ε, υποχρεώσεις από πλευράς των ε, γεωργών, πρασίνισμα και ούτω καθεξής. Εγώ αναρωτιέμαι ποια είναι η βάση στη συνθήκη για όλα αυτά. Γιατί όταν διαβάζει κανείς τη συνθήκη που εξακολουθεί να ισχύει, λέει ότι στόχος της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι η αύξηση της αποδοτικότητας η στήριξη των τιμών κτλ. Αλλά αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας δεν, αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας δεν βασίζεται κάπου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους γεωργούς μας να είναι πιο πράσινοι, να καταπολεμήσουν τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην συνθήκη. Αυτό που κάνουμε εδώ εμείς ε, είναι στην ουσία ότι ξανασυντάσσουμε τη συνθήκη. Εγώ είμαι δικηγόρος ε, και ίσως να ε, είμαι πολύ υπερβολικό συντήρηση της νομοθεσίας, αλλά η συνθήκη είναι μια πράξη στην οποία όλοι θα πρέπει να τηρούμε. Γιατί αυτό που προτείνεται εδώ ξεπερνά το γράμμα της συνθήκης. Ευχαριστώ. Αντιπρόεδρε Βοζιχόφσκι έντονη συζήτηση. Πήραν σύντον όλοι οι παρόντες συνάδελφοι τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Η δουλειά του Λουίς θα είναι πολύ σημαντική. Και τώρα θα ζητήσω από την Κομισιόν να πάρει τον λόγο. Δύο εκπροσώπους της Κομισιόν έχουμε. Πλέβα και Ζούβα. Ποιος θα τα πει πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν στην αρχή αυτής της σημαντικής συζήτησης για το μέλλον του δεύτερου πυλώνα θα ήθελα να πω ότι ο Επίτροπος θα είναι στη διάθεσή σας για να δώσει λεπτομέρειες και τεχνικές πληροφορίες για την πρόταση. Με χαρά άκουσα επίσης ότι σε πολλά θέματα υπάρχει μεγάλη σύγκληση ανάμεσα στην πρόταση της Κομισιόν και την γνωμοδότηση, ε, την γνώμη μάλλον των μελών της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις και μετά θα ήθελα να ζητήσω από τον συνάδελφο Ζωζεφ Σουβαούβα να απαντήσει στις υπόλοιπες παρατηρήσεις. Το πρώτο αφορά την κατανομή των κονδυλίων του δεύτερου πυλώνα. Θα ήθελα να αναφέρω ότι σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής η κατανομή του κονδυλίο του δεύτερου πυλώνα θα πρέπει να γίνει επί τη βάση αντικειμενικών κριτηρίων και προηγούμενων επιδόσεων, δηλαδή τη σημερινή κατανομή κονδυλίων ανάμεσα στα κρατημέλη. Τα αντικειμενικά κριτήρια αναγράφονται στην αξιολόγηση αντικτύπου, για παράδειγμα η ανταγωνιστικότητα, δείκτες όπως η γεωγραφική περιοχή, η απασχόληση, η παραγωγικότητα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επίσης, κριτήρια βιωσιμότητας ή περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, το Natura 2000, τα δάση, τα μόνιμα βοσκοτόπια. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αναφέρω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το θέμα της συνοχής καθώς και ο πληθυσμός. Ε, έγινε ένα σχόλιο σε σχέση με το πώς θα χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα χρήματα ε, για το δεύτερο πυλώνα και πώς θα διευκολυνθεί η χρήση αυτών των ποσών για αποτελεσματική χρήση από πλευρά των κρατών μελών και των γεωργών. Ιδιαίτερα το θέμα της συγχρηματοδότησης είναι αυτό που αναφέρθηκε. Για τη συγχρηματοδότηση θα έλεγα ότι είναι προς το συμφέρον της Κομισιόν να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Και γι' αυτό θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα καταρχήν στις περιοχές που τα χρειάζονται και πιο πολύ. Γι' αυτό και προτείνουμε ένα ψηλότερο επίπεδο συγχρηματοδότησης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, 85% σε σχέση με το 50% ε, για τις υπόλοιπες ε, περιφέρειες. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς θα θέλαμε να διευκολύνουμε τη χρήση των χρημάτων. Αλλά επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η συγχρηματοδότηση δεν μπορεί να αποφευθεί στο πλαίσιο της επικουρικότητας και της κοινή διαχείρισης, shared management. Η συμβολή των δικαιούχων είναι επίσης σημαντική για την ε, Ε, προς χάρη της διαφάνειας Επίσης προτείνουμε άλλες λύσεις για όσον αφορά την χρήση των χρημάτων. Σήμερα δεν υπάρχουν διατάξεις για την ε, ε, εκχώρηση χρημάτων από το Ταμείο Συνοχής επί τη βάση του απλοποιημένου κόστους οι επιχορηγήσεις ε, ε, καταβάλλονται επί τη βάση τιμολογίων. Με μια μεγάλη απλοποίηση μετά από το 2013 θα είναι δυνατόν να καταβάλλονται οι επιχορηγήσεις επί της εξής βάσεως. Ε, στάνταρ κλίμακα κόστους, καταποκοπή ποσό μέχρι τις 100.000 δημόσιες συμβολής και η χρηματοδότηση του εμπορίου με βάση τα διάφορα ποσοστά των κατηγοριών κόστους. Επιπλέον θα μπορεί κανείς εμερικός να αποσμειωθεί σε άμεσο κόστος με τους εξής τρόπους. Ως ένα ε, καταποκοπή ποσό μέχρι 20% επιλέξιμο του άμεσου κόστους, 50% ή επί τη βάση των εφιστάμενων μεθόδων. Ένα παράδειγμα διευκόλυσης δηλαδή των γεωργών στην ισχύουσα πρόταση, στην ε, παρούσα πρόταση. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά τον καθορισμό των ε, λιγότερο ευνοημένων περιοχών. Έγινε ένα σχετικό ερώτημα σε σχέση με την χρήση νέων χαρτών με τον καθορισμό λιγότερο ευνοημένων περιοχών από πλευρά των κρατών μελών. Για αυτό το θέμα θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται η εργασία και η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη επί τη βάση οκτώ βιοφυσικών κτηρίων προετοιμάζουν ε, χάρτες με νέους ε, ε, με, νέα χαρτογράφηση. Ορισμένοι ήδη έκαναν μια οριστική προσωμείωση και έχουν υποβάλει σχετική πρόταση, αλλά κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει αυτή την εργασία. Κάποια κράτη-μέλη αποφάσισαν μάλιστα να τοποθετήσουν τις, τους νέους, τις νέες περιοχές, ε, τις λιγότερο ευνοημένες στο διαδίκτυο, ενώ κάποια άλλα κράτη-μέλη έχουν δυσκολίες να μοιραστούν αυτά τα προσωρινά αποτελέσματα για πολλούς και διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων είναι και το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Γι' αυτό και συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη και σε συμφωνία με τα κράτη-μέλη που είναι οι ιδιοκτήτες αυτών των εγγράφων και που θα μπορέσουμε να σας τα δείξουμε όταν και αν τα κράτη-μέλη συμφωνήσουν γι' αυτό. Και τώρα θα ήθελα ο συνάδελφος να συμπληρώσει τα σχόλια της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μεταξύ άλλων, παίρνω το λόγο για να πω ότι πολλές από τις ανησυχίες ε, και τα αιτήματα ή ερωτήματα των ε, μελών της Επιτροπής σας είναι ενσωματωμένα στην αρχιτεκτονική της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου. Ετέθε ένα ερώτημα τι είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου τελικά. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η κοινή γεωργική πολιτική περιλαμβάνει τρεις μείζονες στόχους που τους υπηρετούν οι δύο πυλώνες, αν μου επιτρέπετε να τα υπενθυμίσω. Ε, μία βιώσιμη παραγωγή τροφίμων που βοηθά στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και επίσης αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. και ισορροπημένη ανάπτυξη των εδαφών. Αυτοί είναι οι τρεις μεγάλοι στόχοι. Η κοινή γεωργική πολιτική μέσω των δύο πυλώνων προσπαθεί να εκπληρώσει αυτούς τους στόχους. Και βέβαια οι δύο πυλώνες ε, σχετίζονται, συνδέονται άμεσα και ε, πολύ στενά. Πρώτον έχουμε το greening, το πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα με τους μεγάλους στόχους της βιώσιμης διαχείρισης των εδαφών ε, της υπαίθρου στη γεωργική παραγωγή και στην παραγωγή δημόσιων αγαθών. Η προοπτική λοιπόν της κοινωνικής πολιτικής στα γενικότερα πλαίσια της στρατηγικής 2020 είναι άκρο σημαντική. Η κοινωνική πολιτική συνολικά προσπαθεί να ανταποκριθεί στους στόχους της στρατηγικής 2020 και σας υπενθυμίζω συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την καινοτομία, την αλλαγή του κλίματος, την ενέργεια αλλά και δράσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για αύξηση του αγροτικού πληθυσμού. Κυρίως βέβαια στοχεύουμε τους νεαρούς αγρότες, κάτι που αναφέρατε και πολλοί από εσάς. Επίσης, μία από τις έξι προτεραιότητες έχει ως στόχο Έτσι φιλοδοξούμε τουλάχιστον να μειώσουμε τον αποκλεισμό και να καταπολεμήσουμε την ανεργία στις αγροτικές περιοχές. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε αυτούς τους δύο πυλώνες ε, για να ανταποκριθούμε στους στόχους της ε, κοινή γεωργική πολιτική. Μίλησε για τον πρώτο πυλώνα. Για το δεύτερο πυλώνα έχουμε και άλλα ταμεία και άλλα κονδύλια που ε, καλούνται όπως και το δικό μας να ανταποκριθούν σε θεματικούς στόχους οι οποίοι ευθυγραμμίζονται άμεσα με τις έξι που έχουν επιλεγεί για την πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μεταξύ αυτών την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και τους τρεις περιβαλλοντικούς θεματικούς στόχους και κλιματικούς στόχους. Δηλαδή, οικονομία με μικρή χρήση άνθρακα, αποτελεσματική χρήση επίσης των φυσικών πόρων. Σε σχέση με αυτούς τους τρεις θεματικούς στόχους, θα ήθελα να σας αναφέρω, να σας υπενθυμίσω ότι εκεί εντάσσονται και δύο από τις μας προτεραιότητες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διάσταση. Για να απαντήσω και σε μία παρατήρηση. Πράγματι ότι αυτό εντάσσεται στην βιώσιμη, στην αηφόρο ανάπτυξη. Θέλουμε μία γεωργία βιώσιμη, αηφόρο. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω το ρόλο δύο μέσων, όχι τριών, ε, τρία είναι, αλλά θα σας τονίσω δύο εγώ, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, έχουμε τα πέντε αυτά τα μία, και οι εταιρικές σχέσεις. Στόχος είναι η διασαφήνιση των προτεραιοτήτων, των βασικών προτεραιοτήτων συνολικά των πέντε ταμείων, για να υπάρξει μια μεγαλύτερη δίκευση της αξιοποίησης των πέντε ταμείων για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών, οι οποίες διέπονται από αυτό το πλαίσιο. Είναι δηλαδή αυτό το στρατηγικό πλαίσιο ένας τρόπος απλούστευσης και διασαφήνισης, γιατί συγκεντρώνει βασικούς άξονες, βασικές δράσεις. Και έτσι δίνει μια συνολική εικόνα και όχι από μονομένες μεταξύ τους αποκομμένες δράσεις. Ε, έχουμε ως στόχο και την μεγιστοποίηση της, ε, των ενισχύσεων. Έχουμε λοιπόν το contract partnership που συνενώνει τις διάφορες ε, συμμετοχές και συμβόλες δίνοντάς τους συνεκτικότητα αλλά και εξατομικεύοντάς τες ώστε το κάθε ταμείο με τη συγκεκριμένη φύση ιδιαιτερότητες που έχει να ανταποκριθεί στους στόχους της στρατηγικής 2020 που προανέφερα. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε που αναφέρω αυτά τα στοιχεία αρχιτεκτονική, αλλά νομίζω ότι μα δίνουν τη δυνατότητα να βάλουμε την ε, συζήτηση αυτή στο σωστό πλαίσιο. Για να μην ε, την αντιλαμβανόμαστε την, πολιτική, την κοινή πολιτική ω ένα πάζελ <laughs> τελείω κατακαιρματισμένη δηλαδή με τι 20 και χθε 40 διαφορετικέ πολιτικέ. Αντίθετα, είναι ένα πλαίσιο διαρθρωμένο που αποτελείται από προτεραιότητε άλλες cross-cutting, όπως είναι η καινοτομία, εγκάρσιες. Έχουμε και την αλλαγή του κλίματος που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και υπάρχουν και μείζονες ανησυχίες, όπως παραδείγματο χάρη με το στοιχείο της καινοτομίας να δώσουμε δυναμική σε όλες τις προτεραιότητες τις οποίες προνέφερα. Με το μέσο της καινοτομία λοιπόν θέλουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε να οργανωθεί με νέο τρόπο η τροφική αλυσίδα, θέλουμε επίσης να προωθήσουμε την τοπική ανάπτυξη. Και δεν αναφέρω τις προτεραιότητες που έχουμε να κάνουμε το κλίμα και το περιβάλλον, γιατί ήδη ε, τα προανέφερα τα σχετικά. Τώρα, αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να απαντήσω στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Πλην αυτών βέβαια για τα οποία απάντησε ο συνάδελφός μου προηγουμένως. Θέλω να αναφερθώ σε μία παράμετρο σε σχέση με, την, ε, με αυτό το αποθεματικό επιδόσεων, απόδοση του 5% που ανέφεραν αρκετοί από εσάς. Αυτό είναι ένα μέσον το οποίο αποσκοπεί αρχικά στα κράτη-μέλη να διατηρηθεί το 5% ε, του φακέλου, του ποσού για κάθε πρόγραμμα. Αυτό το 5% στη συνέχεια πιο καθυστερημένα θα διατεθεί αφού πρώτα έχουν μελετηθεί τα δεδομένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016 σε σχέση με την έναρξη του προγράμματος. Όταν μεταφτάσουμε στο 2019, τότε εκεί πράγματι μπορούμε να επαληθεύσουμε στο πλαίσιο ενός προγράμματος ποιες είναι οι πιο αποδοτικές προτεραιότητες που είχαμε τις καλύτερες επιδόσεις δηλαδή. Και συνέχεια θέλω να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κινδύνων, πράγματι εμείς δεν πληρώνουμε τη συγκρότηση αυτή του, του ταμείου, γιατί ο προγραμματισμός έχει ως βάση μια στρατηγική με επιλογή προτεραιοτήτων. Και στο πλαίσιο της ευελιξίας που έχουν ζητήσει επίσης διάφοροι, μπορούμε να επιλέξουμε τις πλέον κατάλληλες προτεραιότητες για τη στρατηγική η οποία προκύπτει από μία ανάλυση ή τέλος πάντων οι προτεραιότητες που έχουν επιλέγει από τα κρατη Θα πρέπει βέβαια αυτό το δημοσιονομικό φάκελο, το ποσό το που έχει διατηθεί, θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε για να καλυφθούν όλες οι προτεραιότητες που θα έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος στο πλαίσιο της στρατηγικής του. Εμείς λοιπόν με αυτά τα κονδύλια ζητούμε από τα κράτη-μέλη να κάνουν στόχευση, ε, στοχοθέτηση των προτεραιοτήτων. Γιατί αν επικεντρωθούν σε ένα μόνο μέτρο, ίσως κάποια άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να, έχουν, ε, να αποδώσουν και να αποφέρουν αποτελέσματα, δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν. Δεν καλύπτουμε την ε, γεωργοδιατροφική βιομηχανία. Επικεντρωνόμαστε στη Γεωργία, ναι, πράγματι. Και πολύ σωστά, το άρθρο 18 προβλέπει στήριξη σε μέτρα εμπορίας και υπάρχουν επενδύσεις για το τομέα της μεταποίησης βέβαια πράγματι υπάρχει μια προσπάθεια συγκέντρωσης των προσπαθειών προς την γεωργία και όχι προς τη μεταποίηση. Επίσης, υποστήριξη στην καινοτομία, μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερη στήριξη της καινοτομίας. Πράγματι, έχουμε με μεταφορά από τον πρώτο πυλώνα στο δεύτερο πυλώνα, με το κάπινγκ, και θα έχουμε 100% χρηματοδότηση πλέον στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα. Η καλή μεταχείριση των ζώων, η ευζοία των ζώων. Αναφέρθηκε και αυτό το θέμα, πράγματι. Θέλουμε να στηρίξουμε την ευζοία των ζώων, αλλά βέβαια και στο πλαίσιο τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα, το greening, πού εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό. Πρώτο ή δεύτερο πυλώνα ό,τι πάει πάνω από το baseline πηγαίνει στο δεύτερο πυλώνα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Και τι είναι baseline, είναι, ξέρετε πολύ καλά, οι υποχρεωτικέ διατάξεις και οι καλές γεωργικές ε, περιβαλλοντικές ε, συνθήκες και ό,τι άλλο αποτελεί την baseline, του πρώτο πυλώνα, τη βάση δηλαδή. de ces exigences de base euh, données par le premier. Αυτά καλύπτονται από τον πρώτο πυλώνα, λοιπόν. Για τις οργανώσεις των παραγωγών και πώς θα αντιμετωπίσουν πώς θα συνδεθούν με τις ομάδες ε, της Ενώσης των Παραγωγών. Θυμίζω ότι όντως στο δεύτερο πυλώνα έχουμε, προβλέπουμε μια ε, αρρωγή στις ε, ενώσεις των παραγωγών. Έτσι χρησιμοποιούμε ομάδες παραγωγών και σύνδεση αυτών με αυτό που προβλέπεται από το άρθρο 36, μέτρα συνεργασίας δηλαδή, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινέ στρατηγικές αγορές, αγοράς, διευρύνοντας το πεδίο της προσφοράς χωρίς να χρειάζεται να βοηθήσουμε τις διαστάσεις που, σε διαστάσεις που μπορεί τελικά να <clears throat> οδηγούσαν σε ένα επιχείρημα του dead weight, ένα επιχείρημα για το οποίο γνωρίζετε ότι το ελεκτικό συνέδριο έχει επιστήσει την προσοχή των θεσμικών οργάνων. Δεν κάλυψα όλα τα σημεία, κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να ολοκληρώσω. Να λίγα λεπτά ακόμα έχετε. Σας ευχαριστώ. Bien. La question euh, des 25%. Το θέμα του 25% δεν αναφέρεται στο κείμενο. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, δεν αναφέρεται στο κείμενο, αλλά καλύπτεται μέσω των ε, προτεραιοτήτων που αναφέρονται ανάμεσα στις 6. Δύο από τις προτεραιότητες που αναφέρονται στις 6. Αντιπεροσωπεύει μια μεγάλη προσπάθεια για τις προτεραιότητες όπου αφιερώνεται η ανάπτυξη ε, υπαίθρου οι ζώνες φυσικού περιορισμένες ε, εντάσσονται στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα και αποτελούν αντικείμενο και μπορεί να αναφέρονται σε ζώνες ορεινές ή σε συγκεκριμένες ζώνες που πάσχουν από ειδικά μειονεκτήματα. Να αναφέρω ότι στα κλιματικά προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του σχεδίου κανονισμού αναφέρεται ότι δίνουμε τη δυνατότητα στο πλαίσιο της έντασης βοήθειας που προβλέπεται στο παράρτημα 5 του κανονισμού δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρξουν υποπρογράμματα αναθέμα τα οποία προβλέπουν τη δυνατότητα να προσφερθούν ενισχύσεις που ξεπερνούν το 20% της ε, συνηθισμένης πρακτικής του 50%. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά για τις ε, λιγότερο ευνοημένες περιοχές, για τις ορεινές περιοχές που προβλέπεται να δοθεί μέσω ειδικών προγραμμάτων ανά θέμα. Θα σταματήσω σε αυτά. Πιστεύω πως τα κάλυψα όλα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ίσως να σας πω μόνο ότι είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας για να συνεχίσουμε και διμερώς με τις συζητήσεις με τα μέλη για να τους δώσουμε όλες τις τεχνικές διευκρινήσεις τις οποίες ίσως να παρέβλεψα αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο εκπροσώπους της Επιτροπής για αυτή την αυθονία στοιχείων. Είναι σημαντικό η Κομισιόν να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ε, τι περί τίνος πρόκειται και να απαντήσει στις ερωτήσεις ε, των μεμονωμένων ε, βουλευτών. Τώρα, Λουίς, εσύ θα πρέπει να συνοψίσεις τα διάφορα ερωτήματα για να πάμε σύντομα και στο τελευταίο σημείο της ημερής διάταξης, γιατί μετά έχουμε και συνεδρίες των συντονιστών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο από αυτή τη συζήτηση γιατί έχουμε από τη μια πλευρά μια καλή πρόταση της Κομισιόν από τεχνικής άποψη. Εγώ θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω την εξαιρετική τεχνική εργασία που έχει γίνει και που διέπει ολόκληρη αυτή την πρόταση. Η αγροτική ανάπτυξη είναι πολύ πιο συγκεκριμένη από ότι οι άμεσες πληρωμές, αλλά υπάρχει αυτό το μεγάλο πολιτικό ζήτημα που πρέπει να λύσουμε που είναι το δημοσιονομικό και ελπίζω με τη συνεργασία των συναδέλφων και πιο συγκεκριμένα με τους σκιώδεις εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων, με τους οποίους θα έχω επαφές τις επόμενες μέρες ατύπως, εξαιρετικά έντονες όμως, με βάση κάποιες προσωμιώσεις που κάνω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια πολύ ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό γιατί νομίζω πως αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα πρέπει να υψώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο με μια συμπαγή και αραγή θέση για να μπορέσουμε να καταστήσουμε δεκτές τις προτάσεις μας. Νομίζω πως για τα πιο σημαντικά θέματα δεν, νομίζω, δεν θα είναι δύσκολο να φτάσουμε στις συμβαστικές λύσεις. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να συζητήσουμε, ε, πολλές, ε, πολλές λεπτομέρειες όπως για παράδειγμα το θέμα των ειδικών ε, προτάσεων γιατί η Κομισιόν απαγορεύει να γίνουν νέες προτάσεις για ε, νέου είδους καλλιέργειες στα παλιά κράτη-μέλη ε, και δεν λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές αλλαγές κτλ. Είμαι όμως βέβαιος πως θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε καλή συμβιβαστική λύση και ευχαριστώ τους συναδέλφους για όλες τις προτάσεις που έκαναν. Τις σημείωσα και θα προσπαθήσω να τις λάβω όλες υπόψη. Ευχαριστώ. Bene, Περνάμε στο τελευταίο σημείο, χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινή γεωρικής πολιτικής. Ε, δίνω αμέσως το λόγο στον Τζοβάνι Λαβία και ε, ελπίζω πως θα μπορέσει να κάνει όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να κάνουμε και τις συνεδρίες των συντονιστών. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να μπορέσουμε να αφήσουμε όσο γίνεται περισσότερο χρόνο στη συζήτηση που νομίζω θα είναι το πιο χρήσιμο στοιχείο για να εμπλουτίσουμε μέσω των παρεμβάσεων τις εργασίες που κάνουμε και που προφανώς έπειτα θα συμπεριλάβουμε στη γραπτή πρόταση έκθεσης που θα σας υποβάλουμε. Η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι Ε, ενέχεται στην ε, χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της μελλοντική κοινή γεωργικής πολιτικής. Η σημασία αυτών των λειτουργιών έγκυται τόσο στον καθορισμό του μηχανισμού ώστε η κοινή γεωρική πολιτική να καταστεί αποτελεσματική και αποδοτική και ε, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικά όρια και το περιεχόμενο που θα αναπτυχθούν στις άλλες τρεις νομοθετικές προτάσεις. Μέχρι στιγμή οι επαφέ που είχα με διαφερόμενου γεωργικού φορεί και με τα θεσμικά όργανα μου επέτρεψαν να εντοπίσω κάποια θέματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά και επί των οποίων συγκλίνουν οι αμφιβολίες και οι ανησυχίες πολλών και επί των οποίων είναι σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας. Δεδομένου ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα περιοριστώ στο να τονίσω κάποια από αυτά τα θέματα, ώστε να δώσω χώρο ε, στην αντιπαράθεση με τους συναδέλφους και να ακούσω τις θέσεις των περισσότερων για να μπορέσω να τη την λάβω υπόψη στο έγγραφο που θα σας υποβάλω. Το πρώτο θέμα δεν μπορεί παρά να αφορά την χρηματοδότηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Τόσο όσον αφορά το κονδύλια που θα χρησιμοποιηθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο, όσο και οι μηχανισμοί που θα διέπουν την κατανομή των πόρων σε σχέση με το ευρύτερο σενάριο προπολογισμού που ακόμα είναι υποκαθορισμό για την περίοδο 2014 με 2020. Οι αρχικές ανησυχίες αφορούν όντως το χρονοδιάγραμμα έγκρισης του δημοσιονομικού πλαισίου και τα κονδύλια που θα αφιερωθούν στην κοινή γεωργική πολιτική που δεν θα μπορούν παρά να επηρεάσουν το περιεχόμενο της ίδιας της πολιτικής, καθώς ε, οι ίδιοι πόροι συνδέονται άμεσα με τις ε, δεσμεύσεις ε, τις οποίες θα χρειαστεί έπειτα οι γεωργοί να διατηρήσουν και να σεβαστούν καθ' όλη την προγραμματική περίοδο. Ένα δεύτερο θέμα που νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε και να θέσουμε στη σε ευρύτερο προβληματισμό είναι η συνεννόηση ανάμεσα στο Συμβούλιο και την Κομισιόν που ήδη αναφέρεται στην προηγούμενη νομοθεσία ε, όσον αφορά την προσαρμογή στη συνθήκη της Λισαβόνα, την ευθυγράμμιση όπως αποκαλείται και το ρόλο της δυνατότητας ε, εξαίρεσης και παρακολούθησης της Κομισιόν. Μέχρι ότου να καθοριστεί και να βρεθεί μια συμφωνία για την ευθυγράμμιση, τα ίδια θέματα θα προκύπτουν διαρκώς στις νέες διαπραγματεύσεις και τη νέα νομοθεσία που πρέπει να εξετάσουμε και θα καθιστούν πιο περίπλοκη και δύσκολη την έγκριση της ίδιας αυτής της νομοθεσίας, της νέας νομοθεσίας. Άρα λοιπόν είναι να πω να ευχόμαστε ότι θα να μπορέσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα να κλείσουμε τον φάκελο που αφορά την ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε πιο σύντομα στα υπόλοιπα σημεία. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω. Να σας θυμίσω ότι στο θέμα το οποίο πέρασε από αυτή την Επιτροπή και από την Ολομέλεια σε σχέση με την ευθυγράμμιση στη συνθήκη, αυτή η Επιτροπή ήδη είχε εκφράσει κάποιες θέσεις τις οποίες ε, δεν βρίσκουμε στη νέα νομοθετική πρόταση. Αναφέρομαι σε ένα θέμα που εκρεμεί ακόμα στην ε, συζήτηση για την ευθυγράμμιση και αφορά την αποδέσμευση κάποιων χωρών που έχουν ε, περιφερειακό χαρακτήρα στη διαχείριση των πολιτικών ε, ανάπτυξης της υπαίθρου. Είχαμε ζητήσει να υπάρχει μια υποχρέωση όχι, μόνο, όχι πλέον αναπρόγραμμα αλλά σε εθνική βάση. Ενώ σε αυτή την πρόταση προτείνεται εκ νέου η θέση που περιλαμβανόταν στον παλιό κανονισμό πριν την ευθυγράμμιση και πριν από την απόφαση του Κοινοβουλίου. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ε, αφορά το ρόλο τη, αλλά και τη διάταξη των οργανισμών πληρωμής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορικά με αυτό το θέμα ζητήσαμε καθώς η κατάσταση είναι πολύ διαφοροποιημένη, διαφορετική στις διάφορες χώρες. Ορισμένοι έχουν ε, περιφερειακή δίκηση, ενώ άλλοι έχουν εθνικού επίπεδου δίκηση. Ζητήσαμε λοιπόν από την ε, Επιτροπή να μας ε, δώσει ένα σύντομο συνοπτικό πλαίσιο για τις 81 υπηρεσίες και οργανισμούς που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με διαφορετικές βεβαίω καταστάσεις από χώρα σε χώρα ε, για τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην συνταγματική δομή και τις επιλογές που έχουν, σε οποίες έχουν προβεί τα κρατημέλη. Τώρα, σε σχέση με τη διαχείριση του ελέγχου. Και εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει κάποια ε, εμβάθυνση σε σχέση με τις κυρώσεις και με το βαθμό αυστηρότητας των κυρώσεων. Με άλλα λόγια, πρέπει να διευκρινιστεί η σχέση του επίπεδου παράβασης αν αυτό θα πρέπει να σημάνει την πλήρη απώλεια της ενίσχυσης είτε, ή αν θα πρέπει να πάμε σε ένα επίπεδο κυρώσεων ψηλότερο από την ίδια τη βοήθεια που έχει δοθεί. Με άλλα λόγια, αν ένας ε, δεν σεβαστεί απόλυτα του όρου του πρασινίσματο. Θα χάσει μόνο τη βοήθεια που σχετίζεται με το πρασίνισμα ή θα μπορούσε να χάσει και περισσότερα. Και έπειτα έχουμε και τις ε, συμβουλές ε, προς τις επιχειρήσεις όπου υπάρχουν ε, πολλές απορίες. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει ένα κίνδυνο κατάχρηση η χρήση μιας μονάδας πληρωμών να πληρώνει 1500 ευρώ κάθε φορά χωρίς περιορισμούς για την επιχείρηση ή θα μπορούσε κάτι τέτοιο να χρησιμοποιηθεί και με στρεβλωμένο τρόπο και από αυτού φυσικά ζητώ τη γνώμη των συναδέλφων. Έχουμε το θέμα των όρων που θα καθοριστεί από τις επιλογές τις οποίες θα προβούμε. Και έπειτα ένα εγκάρσιο θέμα, το οποίο έχουμε ακούσει πολλές φορές, επανελειμμένος, μια μεγάλη προσπάθεια προς την απλοποίηση. Αλλά αλλά έχω την εντύπωση πως δεν έχουν γίνει και πολλά προς αυτή την κατεύθυνση σε αυτόν τον προτινόμενο κανονισμό που σε πολλά θέματα προτείνει εκ νέου τα όσα είδα υπήρχαν στην παλιά νομοθεσία. Αυτή η απλοποίηση είναι ένα ζήτημα το οποίο επανειλημμένως ζητούν οι γεωργοί και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μπλεκόμενοι φορείς το υπογραμμίζουν για να έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική αποτελεσματική που θα μπορέσει να δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει μια επιπλέον προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Bene, grazie Giovanni. Ε, Σας ευχαριστώ Giovanni. Να ρωτήσω αμέσως τους συναδέλφους αν θέλω να παρέμβουν. Ο Λουίς Καπούλα Σάντος και μετά ο Διευθυντής Μέγκελ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα κανονισμό εξαιρετικά σημαντικό. Ένα κανονισμό που αφορά τη μόνιμη μας ε, ε, ε, ενασχόληση με τη λιτότητα, με την απλοποίηση, τη διαφάνεια, την εικόνα που δίνουμε στους πολίτες για το πώς χειρίζεται το δημόσιο χρήμα η Κομισιόν και άρα ε, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά από πλευρά του εισηγητή μα και εγώ προσωπικά αλλά και από πλευρά τη πολιτική μου ομάδα θα τον διαβεβαιώνω για την πλήρη μα συνεργασία ώστε η δουλειά του να είναι θετική και συνενετική. Bene, grazie Luis. Allora, direttore Ευχαριστούμε. Ο ε, κύριος Μπέγκελε έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Λαβία για νομίζω την πολύ καλή σύνοψη των ε, θεμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση της Κομισιόν για τον οριζόντιο κανονισμό. Πολύ σύντομα θα αναφερθώ στα σημεία που αναφέρατε και θα προσπαθήσω να σας δώσω κάποιες διευκρινήσεις. Αναφερθήκατε στο γεγονός ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στις ε, αποφάσεις ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον κανονισμό αυτών. Γενικά υπάρχει σχέση ανάμεσα στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και όλες τις προτάσεις του κανονισμού που γίνονται, αλλά ειδικά σε αυτή την περίπτωση του οριζόντιου κανονισμού, η σχέση αυτή είναι μάλλον χαλαρή. Ο κανονισμός εξυπηρετεί ώστε να θέσει τους κανόνες σχετικά με το πώς θα διατεθούν τα χρήματα με κανέναν τρόπο όμως ε, δεν λέει πόσα χρήματα θα πρέπει να διατεθούν. Γι' αυτό νομίζω ότι μπορεί ήσυχα να μην συζητάει κανείς ε, τον ε, κανονισμό αυτό χωρίς να φοβάται ότι θα δημιουργηθεί προηγούμενο, διότι ο κανονισμός αυτός θα λειτουργήσει ε, άσχετα από το αποτέλεσμα των ε, διαπραγματεύσεων ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ένα θέμα που μας, που μας απασχολεί και μας ανησυχεί εδώ και κάποιο καιρό είναι ότι μετά την Λισαβόνα έχουμε ε, προχωρήσει σε νέους τόπου. Ε, θα ήταν ωραίο πάντω εάν ε, τα θέματα του κανονισμού 1290 μπορούν να ξεκαθαριστούν. Έχουμε ένα οριζόντιο πακέτο, προ, προβλέπεται ένα οριζόντιο πακέτο, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι, οι σχετικές συζητήσεις. Αναφέρατε Ε, αναφέρατε επίσης ε, μία πολύ ενδιαφέρουσα διαπίστωση. Είχα, ε, είχα, όσον αφορά την ευθυγράμμιση που αναφέρατε, Όσον αφορά λοιπόν την ευθυγράμμιση φαίνεται να υπάρχει μια τροποποίηση και της θέσης του Κοινοβουλίου. Αναφερθήκατε στο θέμα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Τα κράτη-μέλη ε, που έχουν περιφερειακά προγράμματα. Αυτό είναι κάτι που συζητιέται στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Συζητιέται και στα πλαίσια της ευθυγράμμισης. Πράγματι, το Κοινοβούλιο έχει λάβει αποφάσεις τροποποίησης ε, σχετικά με τον κανονισμό 1290 2005. Η Κομισιόν θεωρεί ότι πρέπει να ξεκαθαραστεί το θέμα αυτό στα πλαίσια του κανονισμού για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Υπάρχουν εδώ διάφορες ιδέες, οι οποίες ε, και εξαιτία της δύσκολης συζήτησης για την ευθυγράμμιση δεν έχουν προχωρήσει, αλλά έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις αυτές όσον αφορά ε, τα ε, διάφορα νούμερα. Συμφωνώ μαζί σας, η Κομισιόν θέλει σύντομα ε, μείωση τους ε, μέσω από την διάρθρωση διαφόρων κρατών μελών, ιδιαίτερα τριών, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, ε, που αντιπροσωπεύουν το μισό των σημείων πληρωμών. Ε, είναι πολύ δύσκολο ε, να παρέμβουμε στις δομές αυτές. Τα κράτη-μέλη είναι κατά. Εμείς όμως θα θέλαμε να υπάρξει συγχώνευση κάποιων σημείων πληρωμών σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το έχουμε συμπεριλάβει και στην πρότασή μας. Κάτι ε, τέτοιο θα οδηγήσει σε μείωση των ε, σημείων πληρωμών από 81 ε, σε 74. Οι σχετικές προτάσεις ε, προετοιμάζονται και θα τις ελάβετε στο εγγύς μέλλον. Αναφερθήκατε στο θέμα των κυρώσεων, ε, αναφερθήκατε και στο greening, το πρασίνισμα. Δεν ε, νομίζω ότι πρέπει να εμβαθύνω στο θέμα αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε και τον, ε, σχετικό χρόνο, δεν έχουμε και τον απαραίτητο χρόνο. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η πρόταση του οριζοντίου κανονισμού λέει ότι οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται θα πρέπει να είναι αναλογικές. δεν επιτρέπεται να είναι δυσανάλογες ως προς τις παραβάσεις. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί όμως αναλυτικά όσον αφορά το ε, σύστημα συμβουλών ε, για τους γεωργούς. Εδώ ε, αναφέρατε το θέμα των, των μέγιστων ποσών, 150 ευρώ για την παροχή συμβουλών. Αυτό όμως έχει να κάνει με την ανάπτυξη της υπαίθρου, όχι με τη γεωργία. Ε, θα πρέπει να συζητηθούν αυτά τα ανώτατα όρια και θα πρέπει να εξεταστεί εφόσον δεσμευτούν τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα συγκεκριμένα ποσά, όλο αυτό θα πρέπει να γίνει ε, στα πλαίσια του, της ανάπτυξης της Πέθρου, διότι εδώ αναφέρονται ε, τα ποσά αυτά. Η ε, πολλαπλή συμμόρφωση, το cross compliance είναι ένα σημαντικό θέμα, θα πρέπει να το συστήσουμε όμως ε, ε, κάποια άλλη στιγμή και επίσης όσον αφορά το οριζόντιο θέμα που αναφέρατε, την απλοποίηση. Πράγματι, ο Επίτροπος Τσιόλος επανειλημμένα έχει αναφερθεί στην απλοποίηση που αποτελεί στόχο και της Κομισιόν να απλοποιηθούν, δηλαδή στο βαθμό που είναι δυνατόν οι κανόνες, αλλά θα πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε τον πολιτικό στόχο, πράγμα που είναι αντικείμενο της πολιτικής συζήτησης και εδώ στο Κοινοβούλιο και κατόπιν θα πρέπει να εξετάσουμε ε, οι πολιτικοί στόχοι που θέλουμε, πώς μπορούν να ε, εφαρμοστούν με τον πιο απλό τρόπο. Ο οριζόντιος κανονισμός, όπως έχει προταθεί, περιέχει μια σειρά προτάσεων που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην απλοποίηση, να αναφέρω μόνο τον, την διάταξη που επιτρέπει στα κράτη-μέλη τους ε, ελέγχους επιτόπου να τους μειώσει από 5% σε χαμηλότερο ποσοστό εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι το σύστημα ελέγχου που χρησιμοποιούν λειτουργεί καλά και ότι παράγουν μόνο ε, ελάχιστο περιθώριο λάθους. τα κέντρα πιστοποίησης ε, έτσι μπορούν ε, να ε, οδηγηθούν σε απλοποίηση της λειτουργίας τους, όπως και των σημείων πληρωμών. Επίσης, αναφέρατε ότι οι γεωργοί δικαίως μπορούν να περιμένουν να μειωθεί το διοικητικό, ο διοικητικός φόρτος τους. Αυτό είναι σωστό. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει στα πλαίσια της συζήτησης ε, για τον οριζόντιο κανονισμό, διότι έχει κυρίως να κάνει με την ε, διαχείριση της γεωργικής πολιτικής από τις εθνικές διοικήσεις. Το θέμα του σε τι βαθμό οι γεωργοί ε, πόσο μεγάλο διοικητικό φόρτο έχουν, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στα πλαίσια της ανάπτυξης υπαίθρου και, στις, και στην κοινή οργάνωση αγοράς. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν από ε, μπορούν να ε, συζητηθούν ε, περαιτέρω. Η Κομισιόν είναι πάντα διατεθειμένη να σας ε, παράσχει όλες τις εξηγήσεις, διευκρινήσεις, πληροφορίες και να σας διαθέσει τα απαραίτητα έγγραφα για να σας δείξει καθαρά ποιοι είναι οι σκοποί της πρότασης αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Bene, Ευχαριστούμε, Δόκτωρ Μέγκελ. Γιωβάνι, θες να πεις κάτι συμπερασματικά. Όχι, ευχαριστώ μόνο την Κομισιόν για την ε, διαθεσιμότητά της και εύχομαι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ευθυγράμμισης στη συνθήκη της Λισαβόνας πριν να μπούμε στην ουσία του ζητήματος. Γιατί πιστεύω πως Κάτι τέτοιο θα απλοποιούσε τη δουλειά και θα διευκόλυνε και την επίτευξη των στόχων. Τώρα, ε, σε σχέση με την απλοποίηση, συμφωνώ βεβαίω με την θέση τη Κομισιόν και με τον Επίτροπο ότι είναι ένα από τα στοιχεία κλειδιά και από αυτού πιστεύω ότι έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας. Ευχαριστούμε Τζοβάνι. Ολοκληρώνεται έτσι η συνεδρία της Επιτροπής μας. Ε, να σας θυμίσω ότι η επόμενη μας ε, συνεδρίαση προβλέπεται για τις 28 και 29 Φεβρουαρίου στις 3 το μεσημέρι της 28 Φεβρουαρίου. Παρακαλώ τους συντονιστές να παραμείνουν ε, στην αίθουσα γιατί αμέσως θα ξεκινήσει η συνεδρία των συντονιστών και καλό βράδυ σε όλους τους άλλους. Τέλος συνεδρίασης. Μάρια.